Uh, ladies and gentlemen, I think um, I see you all spread out in this vast chamber, but uh, very well welcome. we We'd be delighted. Um, I know we have a few. Καλημέρα σας. Έχουμε κάποιους ε, εξέχοντες καλεσμένους που κάθονται εκεί άκρη-άκρη. Εάν θέλετε, εάν, μιλώ στους προσκεκλημένους μας, εάν θέλετε να έχετε πιο άμεση συμμετοχή, ελάτε, μπορεί να πλησιάσετε. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ είμαι, σας κουνάω το χέρι, ελάτε, ελάτε. To um, come and join our more intimate circle, um, let me put it that way. Um, uh, Well, good morning everybody. Uh, welcome to um, a uh, session. Καλημέρα σας. Ξεκινούμε αυτή μας πρωινή συνεδρίαση. Τώρα τέλο εβδομάδα πολιτικών ομάδων. Έχουμε θέματα σημερισία ημερησία διάταξη. Πρώτα-πρώτα συνεχίσουμε την σημαντική μα συζήτηση όσον αφορά τι τροπολογίε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ε, το έγγραφο για την δικαιώματα των καταναλωτών και το σχετικό νομοθέτημα. Στι 10.30 θα έρθει ο Επίτροπο ο κ. Σταγιάννη και θα συζητήσουμε για το νομοθετικό πρόγραμμα 2010 2011. Στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε διαρθρωμένος διάλογος Κομισιών Κοινοβουλίου. Τον είδα χτες, χθες το απόγευμα και περιμένει πώς και πώς να έρθει εδώ και να μας πει το, το διάφορα σημαντικά που έχει να μας εξηγήσει πολύ στενή συνεργασία μας με τον κύριο Ταγιάννη έχει το χαρτοφυλάκιο για επιχειρηματικότητα και βιομηχανία. Αυτά όσον αφορά τις ε, ε, αρχικές παρατηρήσεις και σας υπενθυμίζω ότι έχουμε έκτακτη συνεδρίαση Δευτέρα το απόγευμα στις 7 και 4 το και 4 στο Στρασβούργο. Οπότε και θα συζητήσουμε τα της δεύτερης ανάγνωσης για τους κανονισμούς που αφορούν τα υλικά κατασκευών. Σας υπενθυμίζω ότι μεταδίδεται ε, στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Ε, υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στο ημικύκλιο των αδεκασιών θέσεων. Φυσικά δύσκολο να το γεμίσουμε. Έχει 800 Θέσεις υπενθυμίζω. Επομένως, για να δούμε τώρα τι θέματα έχουμε σήμερα. Να πούμε δύο-τρία θεματάκια πριν αρχίσουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατόπιν αιτήματος του εισηγητού να μας ενημερώσει όσον αφορά τις τροπολογίες. Ε, οπότε υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο το οποίο έχετε λάβει. Και σύμφωνα με τη διάταξη, ο κύριος Πέτρη από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίο εδώ βρίσκεται στην αίθουσα, να του σηκώνει το χέρι του, πρόκειται να μας μιλήσει. Και θα συζητήσουμε από αυτό που έχει να μας πει. Επίση, έχουμε την εναρμόνιση διαφόρων διατάξεων για τους καταναλωτές και προχωρούμε στην εξέταση των τροπολογιών όλα αυτά μέχρι τις 10 και μισή. Ε, ο συγητής τώρα, ο κύριος Σουάμπ, μήπως έχει κάτι να μας πει ή να πάμε κατευθείαν ε, στην εισήγηση της Επιτροπής. Καλώς ορίσατε συνάδελφε. Κύριε Πέτρη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ευκαιρία σήμερα που ήρθα εδώ να σας πω μερικές ε, λεπτομέρειες που αφορούν την έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Ιδιώτη μας ζητήσατε να εξετάσουν τις ε, αλλαγές όπως προτείνονται στο σχέδιο του κειμένου για να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε την έκθεση των επιπτώσεων που αφορά την αρχική μας πρόταση επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε με τη μεθοδολογία που έχουμε για την ε, αρχική έκθεση επιπτώσεων. Μελετήσαμε το κείμενο του κυρίου Σβάμ και είδαμε ότι έχουν γίνει 11 σημαντικές αλλαγές. Οπότε προσπαθήσαμε να δούμε τι, τι, τι συμβαίνει, τι άλλαξε σε σχέση με την αρχική μας μελέτη επιπτώσεων. Επίσης, εξετάσαμε αυτές τις αλλαγές σε σχέση με τις ε, ε, τέσσερις αλλαγές στην πολιτική μας που περιέχει αρχική πρόταση. Για να δούμε κατά πόσο με αυτές τις αλλαγές θα λειτουργεί καλύτερη ιστορική αγορά. Επίσης, μελετήσαμε τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών όσον αφορά την ε, νομοθεσία για τις επιχειρήσεις. Τρίτον, τι γίνεται αν έχει βελτιωθεί η νομοθεσία, η κοινωτική και η εθνική με αυτές τις αλλαγές. Τέταρτον, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών όσον αφορά την ε, καταναλωτική, την εμπιστοσύνη του καταναλωτού τέλος πάντων. Και βλέποντας αυτές τις αλλαγές τις 11 μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια ότι μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Έτσι έχουμε πιο στοχοθετημένη και πληρέστερη εναρμόνιση. Αυτέ τι αλλαγέ επίσης. Υπάρχουν κάποιες αλλαγέ που έγιναν για να προστατεύεται καλύτερα ο καταναλωτή, Καλύτερα σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι έγιναν και κάποιες αλλαγέ που έχουν στόχο την αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής του νομοθετήματος. Πρώτα πρώτα όσον αφορά την πιο στοχευμένη εναρμόνιση. Κάτι που όπως ξέρετε είναι και ένα από τα βασικά θέματα της έκθεσής σας. To be excluded from, uh, from full harmonization, uh, for instance the... Μιλούμε για κάποια ενδικά μέσα, ε, κάποια, ε, κάποια μέσα που διαθέτει το καταναλωτής όσον αφορά τις συναλλαγές και ε, άλλους τρόπους για να προστατευτεί. Επίσης έχουμε και κάποιους άλλους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση, την πληροφόρηση του καταναλωτή σε σχέση με κάποιες εξαποστάσεων εξ συμβάσεις και ρυθμίζεται και το θέμα της αναμόνησης των διατάξεων για τις συμβάσεις που συνάπτονται επί τόπου σε κάποιο εμπορικό χώρο. Θεωρούμε ότι έτσι κάπως περιστέλλονται οι φιλοδοξίες της εναρμόνισης. Ε, τώρα έχουμε κάποιο αυξημένο κόστος των συναλλαγών σε σχέση με τη δική μας πρόταση. Ε, πρόκειται για κάποιες διασυνολικές συναλλαγές ε, επί τη βάση το, της εθνικής νομοθεσίας που υπήρχε μέχρι τώρα γιατί σε σχέση με, την, ε, με το δικό μας κείμενο τώρα για να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο. Εναρμόνιση όμως όσον αφορά την εναρμόνιση, όσον αφορά τη συμβάσεις εξαποστάσεως αποστάσεως, αλλά και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την εσωτερική αγορά θέματα τα οποία δεν έχουν περάσει σε εναρμόνιση όπως οι συμβάσεις σε εμπορικό χώρο κατά τη γνώμη μας η συμμόρφωση τώρα απαιτεί δαπάνες από πλευράς των επιχειρήσεων. Απλώς στις δικές αγοράς θεωρούμε ότι είναι αρκετά θετικό το κείμενο του εισηγητού το επίπεδο τρόπο προστασία του καταναλωτή όσον αφορά αυτούς τους τομεί. δεν θα θυγεί από την πρόταση βέβαια όμως από την άλλη μεριά ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αυτές τις αλλαγές σε σχέση με τη δική μας πρόταση μήπως η εμπιστοσύνη του καταναλωτή τώρα ε, μειώνεται σε σχέση με τις διασυνοριακές συναλλαγές γιατί τώρα ίσως θα δημιουργηθεί κάποια σύγχυση στους καταναλωτές. Τέλος, έχουμε τα θέματα αξιολόγηση, τα θέματα κοινοποίηση. Ε, προτείνει εδώ ο εισηγητής να γίνει κάποια ελάχιστη εναρμόνιση. Η ιεραρχία των ενδικών μέσων, η κάποιες εγγυήσεις που παρέχονται από τον, την νομοθεσία, Έχουμε εδώ επίσης επιπλέον ε, υποχρεώσεις για τις ε, κρατικές αρχές αλλά και για την Επιτροπή. Βέβαια, σε, ε, σε αυτό το χώρο τώρα που κινούμε θα είναι δύσκολο να κάτσουμε και να αποτιμήσουμε το, το, κόστος αυτών των επιπλέον υποχρεώσεων των μεν και τον δε και επομένως εδώ δεν μπορούμε ότι έχουμε αποκρισταλώσει άποψη για τις επιπτώσεις ε, των θεμάτων αξιολόγησης, ε, κοινοποίηση, των μηχανισμών αυτών που προτείνεται. Επίσης, όπως προείπα, έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο έκθεσης που οδηγούν στην αύξηση της ε, προστασίας των καταλωτών. Ας πούμε, προτείνεται. Η περίοδος κατά την οποία κανείς μπορεί να καταγγείλει μια σύμβαση πάει στον ένα χρόνο. Επίσης, κάποιο είδους ε, δημοπρασίες μέσω του διαδικτύου και εκεί υπάρχουν κάποιες ε, μεταβολές. Επίσης είπαμε καταγγελία κάποια ε, σύμβαση ή παναχώρηση από σύμβαση για κάποιες αγορές. Ε, σε σχέση με την αποδοχή αυτών των ε, αγαθών που αγοράζονται και πάντοτε μιλούμε για κάποιες συμβάσεις που δεν συναντούνται σε εμπορικό χώρο, σε κατάστημα. Άρα, περισσότερη προσοχή του καταναλωτή τώρα. Επίσης, κάποιες άλλες διατάξεις για την ε, επιστροφή του τιμήματος. Μιλούμε για τιμή πάνω από τα 50 ευρώ οπότε εάν κανείς επιστρέψει αυτά που αγόρασε δεν θα έχει κάποια επιπλέον επιβάρυνση για το κόστος αυτής της επιστροφής των αγαθών. Άρα εδώ τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Μεγαλύτερη προστασία για τον καταναλωτή. Αύξηση του βάρους στις επιχειρήσεις, του κόστου συμμόρφωσης δηλαδή. Η παναχώρηση λοιπόν από τη σύμβαση ε, και σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία, όπου υπάρχει τέτοια νομοθεσία στα κράτη-μέλη, θα επιβαρυνθούν κάπω οι επιχείρησει από την άλλη μεριά. Τώρα, σε πολλέ χώρε μέλη θα προστατεύεται καλύτερο καταναλωτή. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Και άρα, στι χώρε εκείνε ο καταναλωτή θα αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτέ τι συναλλαγέ. Με λίγα λόγια, συνοπτικά, όσον αφορά τι αλλαγέ, έχουμε την πρόσφατη καταναλωτή, ε, από τη μια μεριά επομένω, μεγαλύτερη προστασία, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, αλλά και περισσότερε επιχειρήσει. Αυτό ήταν μια πολιτική επιλογή. Ε, την κάνετε εσεί, ε, θα αποφασίσετε εσεί και το Συμβούλιο σε πολιτικό επίπεδο και τέλος έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές αφορούν τους ορισμούς, αφορούν το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης γιατί εδώ πέρα στο κείμενο προτείνεται η αναθεώρηση του ορισμού που αφορά τη συμβάση εξ Να επανεισαχθεί το ότι θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει τη μορφή της ε, σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως. Αυτό τώρα έχει αλλάξει με την αρχή πρόταση. Σε σχέση λοιπόν με το, το ότι ο αγοραστής ε, έρχεται σε επαφή με τον πολιτή και συμφωνεί κάτι. Αυτό τώρα έχει αλλάξει με την αρχή μας πρόταση. Θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης δεν επιτυγχάνει το ίδιο επίπεδο προστασία του καταναλωτού όπως η δική μας πρόταση. Ούτε θεωρούμε ότι έτσι τα παραθυράκια του νόμου αντιμετωπίζονται όπως τα είχαμε εμείς επισημάνει για τις ε, συμβάσεις εξ Αυτά τα οποία ισχύουν με την... Ε, αυτά τα οποία υπάρχουν τώρα τα κενά στην ισχύουσα οδηγία στις συζητήσεις που έγιναν όλα αυτά έχουν επισημανθεί στο Συμβούλιο και εν κατακλείδη Όλες αυτές οι αλλαγές Έχουμε αυτές τις αλλαγές δεδομένες τώρα και είναι σαφές ότι το κείμενο του εισηγητού μας οδηγεί σε καλύτερη προστασία του καταναλωτή ως προς πολλά. Ε, από την άλλη μεριά. Τώρα, έχουμε μία ελάχιστη εναρμόνιση σε διάφορους τομείς. Ε, και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κατάτμιση της προστασία του καταναλωτή αλλού υπάρχει, αλλού δεν υπάρχει, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο οπότε αυτού του είδου η στοχευμένη εναρμόνιση οδηγεί στο ότι οι καταναλωτές δεν θα φερθούν την ενιαία εσωτερική αγορά τόσο όσο με τη δική μας πρόταση. Παρ' όλα αυτά, που είναι το σημαντικό, Υπάρχει ένα αντιστάθμιο, ένα αντάλλαγμα με την πρόταση αυτή στα σημεία που υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και η εναρμόνιση τώρα θα στοχεύσει στο να καλύψει τις συμβάσεις εξ και τις συμβάσεις εκτός εμπορικών χώρων. Οπότε Ω προς αυτά τα σημεία θα έχουμε βελτίωση τη λειτουργία τη ε, ενιαία ιστορική αγορά σε σχέση με το τι ισχύει τώρα. Για όλα αυτά που μας είπατε και πραγματικά μας αναλύσατε εξαιρετικά την ε, έκθεση και πιστεύω ότι μας βοήθησατε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τώρα κάποια σχόλια από τους σκιώδεις πριν περάσουμε στη δικιά μας συζήτηση για τις ε, τροπολογίες. Θα δώσω λοιπόν πρώτο το λόγο στον κύριο Σβάμπ να μας πει την άποψή του και μετά τους ε, σκιώδεις ε, να μας πούνε αν έχουν καταφέρει να εξάγουν κάποια συμπεράσματα ή κάποια επιπλέον συμπεράσματα μετά από αυτά που μας είπε η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ε, και ο Πρόεδρος μόλις είπε, και εγώ είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, έκανε τελικά αυτή την εργασία σύγκρισης ε, της επίπτωσης του κειμένου της Επιτροπής και του τροποποιημένου κειμένου, έτσι δηλαδή όπως τροποποιήθηκε από την έκθεση έτσι όπως ε, εξελίχθη η πλειοψηφία ε, μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και ε, συμφωνώ <clears throat> με την Επιτροπή διότι συμφώνησε μαζί μου και με πολλούς συναδέλφους ότι μπορούμε να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να αφαιρέσουμε την ευελιξία της Επιτροπής βέβαια και των κρατών μελών. Ε, βεβαίως ε, όπως εγώ υπέβαλα ή στις ε, τροπολογίες μου χρειάστηκε να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές και άλλωστε ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουν οι συμβάσεις δηλαδή τα οργανωμένα συστήματα διεκπαιρεώσεως να μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες διότι ε, όπως είπε και η Επιτροπή δεν πρέπει να μειώσουμε την προστασία των καταναλωτών και χρειάζεται ενδεχομένως ε, να ε, κάνουμε προσαρμογές όπως απέδειξε υπήρξε η αίτηση για για μία ε, ε, έκθεση ε, αξιολογήσεως των επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει, κυρία Γκέπχαρτ. Λοιπόν, για να ακούσουμε πρώτα όλα τα σχόλια των σκιωδών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά τους συναδέλφους μου θα ήθελα να τους ζητήσω συγγνώμη διότι ο κύριος Χορέα και εγώ γυρίσαμε χθε το βράδυ από την συνεδρία της πολιτικής ομάδας στη Βουδαπέστη για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην πολιτική ομάδα. Οι άλλοι συνάδελφοι έμειναν εκεί οπότε γι' αυτό σήμερα υπάρχει πολύ κακή παρουσία και συμμετοχή της Επιτροπής μας, ασύνηθες ε, δηλαδή. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σκέφτηκε τόσο πολύ τις προτάσεις του εισηγητή και εμείς ε, θέλουμε να γνωρίζουμε ε, τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί ε, κινείται όπως κινείται. Εν πάση περιπτώσει όμως με εκπλήσει ο τρόπος με τον οποίο έγιναν αυτά διότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει είναι μετά από επιθυμία του Κοινοβουλίου και εγώ σας συντονίστρια δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε ζητήσει μια τέτοια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις τροπολογίες των Ευρωβουλευτών. Άρα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω αν λειτουργούμε έτσι τώρα. Αυτό που βρίσκω επίσης προβληματικό και θα ήθελα να διευκρινίσουμε ε, ή στη συζήτηση και θέλω να σας προειδοποιήσω είναι ότι δεν δεν πρέπει να συγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόταση του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κάποια στιγμή ε, κάποιας προτάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αυτό που συζητάμε εδώ στην οδηγία είναι ποια είναι η σύγκριση με τα ισχύοντα δικαιώματα και αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ να μην μπερδέψουμε τα πράγματα και να γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος ομιλούμε. Όταν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτόν τον οποίο ζητά ο εισηγητής αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι ουσιαστική η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αλλάζει για τους πολίτες εάν γίνουν αυτά τα οποία προτείνει ο Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρέπει να ρεχθεί ρητός. Καμία αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα νέο έγγραφο γιατί εγώ δεν προεξοφλώ ούτως ή άλλως ότι όλα αυτά πρόκειται να είναι προς όφελός μας. Αυτό που θέλω επίσης να διευκρινίσω είναι ότι στη διαθεσμική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου ε, και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας αλλά τις αποφάσεις λαμβάνουν το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο και έτσι πρέπει να παραμείνει η κατάσταση. Σήμερα το πρωί όμως είδα ένα χαρτί πάνω στο τραπέζι το οποίο δεν έχω κοιτάξει καν. Είναι ένα αγγλικό έγγραφο άρα δεν μπορώ να το σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει. Ε, αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αυτό το έγγραφο πρέπει να μας πει τι εννοεί με τα συν και τα πλήν και τις ε, επιφυλάξεις διότι εγώ δεν ε, μπόρεσα κοιτάζοντας το να καταλάβω περί τίνος πρόκειται και γι' αυτό δεν μπορώ να αξιολογήσω και το έγγραφο αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι αυτό είχε συζητηθεί τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, κατόπιν πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ και ε, γι' αυτό δεν ε, επηρεάζει βέβαια ή δεν μειώνει τις αρμοδιότητες μας σαν αξιολογητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση για αξιολόγηση μεθόδου και νομίζω ότι με την οδηγία αυτή στην ουσία έχουμε μια κατάρα ε, πάνω από τα κεφάλια μας. Δηλαδή κάθε φορά αρχίζουμε και συζητάμε για όρους, για προϋποθέσεις, τέλος πάντων για περιφερικής σημασίας και ενδιαφέροντος πράγματα. Βεβαίω θεωρώ ότι η εργασία της Επιτροπής είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όπως κάθε ενδιαφέρουσα εργασία είναι και βαθύτατα χρήσιμη και επομένω, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει οποιοδήποτε λόγος να στενοχωρηθούμε ή να λυπηθούμε για αυτά που ακούσαμε. Πέραν τούτων των παρατηρήσεων, ε, πρέπει να πούμε τα εξής. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι παρατηρητής αδέκαστος και αντικειμενικός κριτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρωτοβουλία του κειμένου και μετά αξιολογεί τις τροπολογίες, οι οποίες τροπολογίες προέρχονται από την έκθεση όπως ισχύει εδώ ή αύριο μπορεί να αξιολογήσει τροπολογίες οι οποίες έχουν εκπονηθεί από άλλους, όχι από τον ίδιο τον εισηγητή, όπως μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν μπορεί να είναι και έτσι και αλλιώς ταυτοχρόνως. Δεν μπορεί να είναι δύο πράγματα μαζί. Ε, ε, και νομίζω ότι ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζει, κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν το Κοινοβούλιο και τα οποία ενδεχομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται κτλ. Επίση, είναι σαφέ ότι δεν ε, θέλω να γίνω βασιλικότερο του βασιλέω ε, πάνω στο κείμενο αυτό. Όμω πιστεύω ότι θα πρέπει να το εμβαθύνουμε στοιχείο στοιχείο-αναστοιχείο και βεβαίω προτίθεμαι να το πράξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης νομίζω ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν έλεγα ότι μπορώ να σχολιάσω αυτό το έγγραφο το οποίο δεν έχω διαβάσει. Από τα όσα όμως έχω ακούσει, εκείνο που εγώ καταλαβαίνω είναι η σύγκριση μεταξύ των ε, ε, προστασίας των καταναλωτών των δικαιωμάτων που έχουν σήμερα και πώς αυτά θα αλλάξουν με τις τροπολογίες και την ε, έκθεση τελικά. Επομένως, αυτή είναι η σύγκριση που θα ήθελα να κάνω εν καιρό όταν εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφέστατα κατέδειξε τις απόψεις της. Λοιπόν, κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει επί της εργασίας της Επιτροπής ή θέλετε να ε, ξεκινήσουμε επί της ουσίας της κυρία θέλετε να μιλήσετε για το έγγραφο της Επιτροπής ή να κάνετε κάποια γενικότερα σχόλια για τον κανονισμό γενικότερα σχόλια. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο, να ευχαριστήσω βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε αυτήν την ε, εργασία. Είναι πάντα χρήσιμο να έχουμε εκπροσώπους τη Επιτροπής και να συζητούμε και είναι πολύ χρήσιμο οι εκπρόσωποι τη Επιτροπής να συζητούν με, τους, ε, τον εισηγητή και του κοιόδης εισηγητέ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σφάμπ, έτσι ώστε να ε, εμβαθύνουμε λίγο στην συζήτηση. Έχουμε και ένα έγγραφο από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ενδεχομένως φαντάζομαι το έχετε διαβάσει και θέλετε να εξάγετε κάποια συμπεράσματα ε, από το έγγραφο αυτό. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε μια επικαιροποιημένη άποψη ε, για την φάση στην οποία βρίσκονται οι συζητήσεις, ε, τις επαφές σας με τους σκιώδεις και την κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να κινηθούμε. Uh, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε και για την ψηφοφορία του Δεκεμβρίου. Κύριε Σβάμπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω με τη μελέτη την οποία παρουσίασαν ε, οι δύο καθηγητές ε, για την συνάδελφο Wallis που δυστυχώς δεν παρίσταται σήμερα αλλά συγχρόνως συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Γκέπχαρτ ότι ε, εδώ δεν πρόκειται μόνο για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να δούμε ποια είναι η νομική κατάσταση σήμερα και όσον αφορά την ε, ε, μελέτη την οποία εμείς αναθέσαμε στους δύο καθηγητές ε, προσπαθούμε να την προχωρήσουμε διότι η μελέτη η οποία έγινε για την κυρία Γουόλη στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δείχνει τι μπορεί, πώς μπορεί να προχωρήσουμε. Η μελέτη αυτή έχει γίνει από τους κυρίους Χάουελ και Ράι Βέβαια δεν είναι δυνατόν σε λίγες ε, μέρες ε, να μπορέσει κανείς ε, να καταλήξει εντός ο λίγων ημερών σε, μία τόσο, σε ένα τόσο ειδικό θέμα. Και έτσι δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την έκθεση του καθηγητή Χάουελς, λέγε ότι η περίπτωση Γκίσπρεχτ θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο ε, στις εξελίξεις και ε, επίση όσον αφορά το 2021-2022 ε, βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για ή πλην κυρία Γκέπχαρτ αλλά πρόκειται για τα υπέρ και τα κατά δηλαδή προσπαθεί να συγκρίνει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτές της δικιάς μας αξιολογήσεως και αυτής της κυρίας Γόλης δηλαδή ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη εναρμόνιση και αυτό μας δείχνει ότι ε, στο σχέδιο της εκθέσεώς μου από την αρχή είχε προταθεί ε, μία μεικτή μορφή και ε, εδώ επειδή βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος μετά από την εξέταση ε, των 600 ε, τροπολογιών αγγλικά πρέπει να σας πω ότι τώρα τελειώνει η γερμανική μετάφραση δεν έχω καν κοιτάξει αν υπάρχουν λάθη ή όχι αλλά από το αγγλικό κείμενο βλέπουμε ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και ε, ε, όσον αφορά τι απόψει των διαφόρων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έχουμε μία κοινή θέση και η κοινή θέση, την κοινή θέση αυτή συμμερίζονται και οι υπόλοιποι. Όσον αφορά το άρθρο 5 όπου η γραμματεία απουσιάζει και εύχομαι καλή ανάρρωση στον υπεύθυνο που είναι άρρωστο Βλέπουμε σε σύγκριση με την έκθεση του καθηγητή Ράιχ ότι αν αναφερθούμε και εξαιρέσουμε ορισμένες υπηρεσίες οι υπόλοιπε εξαιρέσει των κρατών μελών για την ασφάλεια και την υγεία ε, καταλήγουν στο ότι μπορούν όλες αυτές οι εξαιρέσεις να συγκεντρωθούν σε ένα κεφάλαιο και βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων διαπιστώνει ότι στα κεφάλαια 2 και 3 έχουν γίνει πρόοδοι όχι μόνο στο θέμα της νομοθεσίας αλλά και στο θέμα της προστασίας των καταναλωτών. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά αυτά τα ε, θέματα της μελέτης και γι' αυτό τώρα ε, θα ήθελα να τοποθετηθώ στις, ε, στα σχόλια των σκιωδών εισηγητών και για να ξέρουμε όλοι πού βρισκόμαστε και να καθορίσουμε τις προθεσμίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Πρώτη φορά συναντηθήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές πριν από δύο εβδομάδες όπου έγινε καταρχήν μία συζήτηση όσον αφορά αφορά τις δυνατότητες συμβιβασμού και δεύτερον διαπιστώσαμε ότι ακόμη δεν είχαν ετοιμαστεί οι μεταφράσεις ακόμη και αν τα κείμενα υπήρχαν αγγλικά είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε αργότερα όταν θα έχουμε τις μεταφράσεις και θα καθορίσουμε και ε, το χρονοδιάγραμμα 23 ε, Νοεμβρίου την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούμε στο Στρασβούργο και θα αρχίσουμε ε, να εξετάζουμε ε, τις ε, δυνατότητες συμβιβασμών στο κεφάλαιο 4 των ε, τροπολογιών και αυτή την εβδομάδα οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων είχαν την πρώτη συνεδρίασή τους, ήδη προετοιμάστηκαν και υπάρχουν ρεαλιστικές καλές προοπτικές για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό παρόλο που το αποτέλεσμα θα διαφανεί στην ψηφοφορία. Όσον αφορά το κεφάλαιο 4, τα ουσιαστικά είναι το άρθρο 26 και 28 στο άρθρο 22 όσον αφορά τις παραδόσεις και την νομιμότητα και τα άλλα θέματα του κεφαλαίου 4 δεν υπάρχουν και τόσες πολλές τροπολογίες και αυτές οι οποίες υπάρχουν ουσιαστικά μπορούν να συμβιβαστούν δηλαδή στο άρθρο 22 πρέπει να δούμε αν πρέπει να υπάρξει μία υποχρεωτική προθεσμία εάν το εμπόρευμα δεν παρεδώσει όσοι έπρεπε ε, σύμφωνα με την τωρινή κατάσταση και ή αν θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η προθεσμία και θα καλυφθεί από την πλήρη εναρμόνιση ε, με το ότι όλοι δεν μπορούν να καταλήξουν στην ίδια λύση αποδεικνύεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όπου όμως μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό χωρίς όμως να πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη ελεύθερα διότι τότε θα μείνουμε στο επίπεδο που έχουμε τώρα. Ε, υπάρχουν και άλλα προβλήματα ότι παραδείγματο χάρη πρέπει να γίνουν ορισμένοι συμβιβασμοί πρέπει να δούμε αν τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα ε, να προβλέψουμε ε, την συνέχεια με την οποία θα προχωρήσουμε ή όχι και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας νομοθεσίας και εφόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε ε, την ε, ελάχιστη εναρμόνιση θέλουμε να αφήσουμε πλήρη ελευθερία στα κράτη αλλά να καλυφθούν και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Και βλέπουμε ότι σε άλλα θέματα έχουμε μια ευρία ποικιλία, σαν μια ανθοδέσμη θα έλεγα. Και υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα, πάρα πολλές προθεσμίες και όσον αφορά ε, τις θέσεις αυτών που ζητούν πλήρη εναρμόνιση και ανθίστανται στις τροπολογίες υπάρχει η δυνατότητα της προθεσμίας τριών ετών συν ένα για επιστροφή αλλά ε, όσοι θέλουν πλήρη εναρμόνιση ε, σκέφτο, κλείνουν προς αυτή τη λύση λύση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι δεν θέλουμε να μειώσουμε το δικαιώματα του καταναλωτών σε κανένα κράτος και εφόσον υπάρχει στην ε, Φιλανδία και αλλού διατάξεις ε, όπου θα μειωνόταν με τις εξελίξεις η μείωση ε, των καταναλωτών. Στη Γερμανία δεν ισχύει το ίδιο διότι παραδείγματος χάρη έχουμε πέντε χρόνια δυνατότητα αναθέσεως αδείας αλλά πάλι ε, υπάρχει μία ε, σαφής διαφοροποίηση μεταξύ της ελάχιστης ε, εναρμονίσεως όπου ορισμένοι συμφωνούν και τις πιο ευξημένης την οποία ζητούμε. Εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από ό,τι υπάρχει τώρα και αυτό θα το συζητήσουμε στις 23 του μηνούς όταν θα συναντηθούν οι συντονιστών. Επίσης δεν ξέρω τι γίνεται με το Συμβούλιο, ίσως θα μπορέσει να μας ενημερώσει ο εκπρόσωπος διότι στις 23 Νοεμβρίου θα συναντηθούμε και μετά και πάλι στις 6 και στις 7 Δεκεμβρίου και αυτό που με στενοχωρεί ήταν ότι στην αρχή είχαμε ε, ζητήσει να συναντηθούμε αν ήταν δυνατόν και στις 24 Νοεμβρίου τα απόγευμα γιατί θα χρειαστούμε πολύ χρόνο για να συντονιστούμε αλλά ε, η Γραμματεία των Επιτροπών ε, μας ζήτησε να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την ημερομηνία για να προωθήσουμε με την νομοθεσία για την ενιαία αγορά και επειδή άλλοι προωθούν και αυτή την νομοθεσία και χρειάζεται χρόνος για την οδηγία ε, με ενδιαφέρει να ξέρω τι ε, λέγουν οι ε, συνάδελφοι δηλαδή μήπως αυτό το σλότ της ενιαίας αγοράς μπορεί να μεταφερθεί στις 23 το απόγευμα αυτά ήθελα να σας πω θέλω να ακούσω τις απόψεις απόψεις των άλλων και προσβλέπω σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την εργασία σε όχι απαραίτητα ενώπιον κοινού, αλλά μεταξύ μας. Ε, ε, και όσον αφορά τον πίνακα, 90-20, νομίζω ότι ε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον πιστεύω θα ήταν να δούμε πώς ε, βλέπουν ε, τα πράγματα και οι διάφοροι σκιώδεις, ε, με ποιο τρόπο δηλαδή αντιμετωπίζουν την εργασία αυτή, τουλάχιστον αυτή τη γραμμή σαν πρόεδρος θα ακολουθήσω στη συζήτηση. Θα κάνουμε τώρα λοιπόν ένα γύρο τραπέζης όλων των σκιωδών εισηγητών. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γκέπχαρτ, μετά έχουμε Ροσφόρ. Δεν ξέρω ποιο θα μιλήσει για τους πράσινους σήμερα. Ο κύριος Μπέλεν είναι εδώ. Ενδεχομένως, ναι. Ωραία, θα κάνουμε λοιπόν ένα γύρο τραπέζι σε των ε, σκιωδών εισηγητών και βεβαίως είναι καλοδεχούμενο όποια σχόλια έχουν και μεμονωμένα μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ δεν με υλώ πιο ε, ευραίος όπως και ο κύριος ρωσοφόρα, αλλά θυμάστε ότι είχε πει η συνάδελφος ότι δεν θα μπορέσει να έρθει ε, γιατί ε, είχε μία σημαντική εκδήλωση δεν θα αναφερθώ τώρα στη μελέτη αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να ακολουθήσω αυτό που είπε κύριος Ροσεφόρ. Δηλαδή να δούμε ε, το περιεχόμενο, να μην μιλάμε ε, ασαφώς διότι τότε δεν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ε, διατυπώσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και εγώ δεν θα κάνω τώρα σχόλια για τις μελέτες. Απλούστατα θα ήθελα να σας πω ότι εγώ έχω διατυπώσει σαν τροπολογίες εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος και τι θεωρώ ότι πρέπει πρέπει να ε, καταστεί σαφές. Καταρχήν δεν θέλουμε πλήρη εναρμόνιση όπως την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ουσιαστικά θέλουμε μία μεικτή μορφή. Ε, όσον αφορά το άρθρο 4 έχουμε υποβάλει ε, μία πρόταση και για το σύνολο επίσης έχουμε διατυπώσει την ελάχιστη εναρμόνιση για να ξέρουμε τι δικαιώματα πρέπει πρέπει να έχουν οι καταναλωτές ε, για να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε και ε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στην πολιτική μας ομάδα και να δούμε πού μπορούμε να δεχθούμε ε, ενδεχομένως μία πλήρη εναρμόνιση σε ορισμένα σημεία. Δεν θα προχωρήσουμε όπως θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όπως άλλωστε πρότεινε και ο κύριος Σφάμπ για τη δική του πολιτική ομάδα για τους σοσιαλδημοκράτες καταρχάς πρόκειται για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό μας απασχολεί και εκεί δεν συμφωνούμε διότι ε, ε, μιλάμε εδώ για μια οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία τους. Πρέπει να υπάρχει αυτή η προστασία και ο στόχος είναι προστασία και όχι εσωτερική αγορά διότι διαφορετικά θα έπρεπε να έχουμε ονομάσει την οδηγία αυτή ε, την ασφάλεια των καταναλωτών και την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου δεν δεν πρέπει να παραμυθιάζουμε τους καταναλωτές και να τους ε, λέμε ότι θα τους πουλήσουμε προστασία των καταναλωτών εάν στην οδηγία υπάρχουν διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία επιζητούμε. Όσον αφορά τα δικαιώματα προς όφελος των καταναλωτών πιστεύω ότι πρέπει να διευρυθούν περισσότερο από ό,τι προβλέπεται εντός των κρατών μελών και αυτό μπορεί να γίνει βαθμιαία. Αυτό ούτως ε, ζητούμε σαν κοινοβούλιο εδώ και 20 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει όλο και περισσότερο σε μία σύγκληση των νομοθεσιών. Γι' αυτό και στα στοιχεία τα οποία έχω και στις, ε, τα μηνύματα που έχω λάβει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να υπάρξει αποτόμως μία πλήρη αλλαγή του ε, συμβατικού δικαίου. Πρέπει ιδίως να προστατεύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους, να μην ε, δηλαδή τους επιβάλλουμε όλα αυτά τα οποία συλλήβδην προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σχετικά με τα μεμονωμένα κεφάλαια. Κεφάλαιο 1. Είναι το κεφάλαιο όπου σαν πολιτικό πολιτική ομάδα μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρξει μία εναρμόνιση για να έχουμε παντού τους ίδιους ορισμούς όσον αφορά τα, τους καταναλωτές, τα δικαιώματά τους και για να αποφιευθούν οι νομικές ασάφειες. Οι μελέτες των καθηγητών Σουλ και Έλκερ δείξαν ότι οι ε, καταναλωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν αυτά τα θέματα, ε, μπορούν να τα διευρύνουν και ως εξ τούτου γι' αυτό διατύπωσα τις προτάσεις και τροπολογίες που διατύπωσα ε, για τις κινήσεις στα κράτη-μέρη. Επίσης επιπλήττουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διότι όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες δεν τις λαμβάνει υπόψη και ξεχνάμε ότι εισάγονται στην αγορά νέα προϊόντα και έχει χαθεί η ευκαιρία να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις σε έναν τομέα που δεν υπάρχει ήδη ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Εκεί θα ήταν χρήσιμο να καταρτιστεί κοινό δίκαιο κατά τρόπο ώστε όλα τα κράτη-μέλη να κινούνται με τον ίδιο τρόπο εφόσον δεν υπάρχει ήδη κάτι στα κράτη-μέλη. Αυτό όμως ε, δεν το χρησιμοποίησε το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε να υπάρξει μία διόρθωση. Επίσης όσον αφορά τον ορισμό των εμπορευμάτων ε, θα ήθελα να ληφθούν υπόψη και τα ψηφιακά προϊόντα δηλαδή ε, την οι πωλήσει του λογισμικού και να διευρύνουμε το εμπορικό δίκαιο διότι έχω και εγώ διαπιστώσει ότι αν πάω στο μέσο του διαδικτύου να αγοράσω ένα γερμανικό ε, ε, ε, ένα γερμανικό λογισμικό και νομίζω το αγόρασα στη Γερμανία και όταν βλέπω ότι μου αφαιρούν και εμβαστικά από το λογαριασμό μου μου αντιλαμβάνουμε ότι ίσως η εταιρεία που μου πώλησε το λογισμικό ήταν π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στη Γερμανία. Ε, αυτά όσον αφορά το α, ε, άρθρο 1. Άρθρο 2 όσον αφορά ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το κεφάλαιο 2 δεν θα έπρεπε να αναφέρεται μόνο στις ευρωπαϊκές ε, ε, υποθέσεις και συναλλαγές και θα πρέπει να το εξαιρέσουμε από την ρύθμιση γιατί πιστεύω ότι το άρθρο 2 και 3 μας δημιουργεί προβλήματα. Το άρθρο 5 δικαίωμα ενημέρωσης ε, θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή κοινή διατύπωση πληροφόρησης, να εξαντλήσουμε εκεί τα κοινά στοιχεία χωρίς να εμποδίσουμε την ευελιξία των κρατών μελών και να μην κλείσουμε την πόρτα στα κράτη-μέλη που θέλουν να νομοθετήσουν εσωτερικά. Να υπάρξει απλώς ένα πλαίσιο όπου θα λέμε, όπως σας είπα και στην τροπολογία μου, ότι μπορούμε να κινηθούμε ασχοληθούμε με ε, διαφορετικούς ευέλικτους τρόπους. Τώρα, όσον αφορά το, τα, επόμενα κεφάλαια το, στο κεφάλαιο 2 θέλουμε ε, να υπάρξουν αλλαγές διότι δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης αλλά ε, θα πρέπει να δούμε δικαίωμα υπαναχώρησης αλλά πώς θα διαμορφωθεί αυτό δηλαδή να λύσουμε και το θέμα των εξόδων που θα συνεπάγεται μία τέτοια ανάκληση ή παναχώρηση. Οπότε πρέπει να υπάρχει μία σαφής διαδικασία η οποία θα είναι εμφανής και άλλωστε ε, το δικαίωμα της ε, αποδείξεως παραμένει εις τον ε, έμπορο και όχι στον καταναλωτή για να μπορεί να ισχύσει το ίδιο που ισχύει τώρα στη Γερμανία Κεφάλαιο 3 ε, όσον αφορά α, τις, ε, συμφωνίες, τις ε, συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά, τα τεχνικά στοιχεία και έχουμε υποβάλει ορισμένες ορισμένες τροπολογίες για την ελάχιστη εναρμόνιση και για την περαιτέρω διεκπαιρέωση αλλά αυτό το οποίο με προβλημάτισε είναι ότι θα πρέπει να, ε, ε, να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορούμε να, κλείσουμε να αποκλείσουμε την εναρμόνιση και δεν ξέρω ε, τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στα 27 κράτη. Εγώ αυτό που μπορώ να κρίνω είναι οι επιπτώσεις στο γερμανικό δίκαιο και όχι στα 27 δίκαια και ήδη είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική όσον αφορά αυτό το σημείο. Για να συντομεύσω, κεφάλαιο 4. Πιστεύω ότι όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις πωλήσεως, εκεί πιστεύω ότι αποκλείεται να υπάρξει ε, πλήρη εναρμόνιση διότι τα εθνικά δίκαια ε, διαφέρουν πάρα πολύ και δεν μπορούν να ενοποιηθούν στα γρήγορα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του τρόπου, πληρωμή ε, του τρόπου πληρωμής που να μην συνεπιφέρει επιπλέον έξοδα και να επιτρέπει και την ε, επιστροφή ε, των χρημάτων. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5, ε, εδώ που ε, αναφερόμαστε ε, στα δικαιώματα των καταναλωτών πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρη εναρμόνιση και δεν νομίζω ότι εδώ πρόκειται να διαφωνήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας και όσον αφορά το κεφάλαιο 6 της Γενικές Διατάξεις πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την επιτροπολογία που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πιστεύουμε ότι δύο πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα των καταναλωτών τα οποία διακυδεύονται και δεν ε, νομίζω ότι είναι κακό να συναποφασίζει εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Αυτά ήταν στα γρήγορα μία σκιαγράφηση των τροπολογιών της πολιτικής μου ομάδος ε, είτε τις δικές μου είτε των ε, συναδέλφων μου ε, εν ονόματι της πολιτικής ομάδες και για να συνοψίσω θεωρούμε ότι η εφαρμογή της ελάχιστης εναρμόνισης έτσι όπως έχει διατυπωθεί μέχρι στιγμής ήταν η σωστή οδός όχι μόνο λόγω της διαφορετικής προστασίας των καταναλωτών καταναλωτών που ισχύει στα κράτη-μέλη όπου δεν μπορεί κανείς ε, να ε, περάσει ε, με, τον ίδιο τρόπο και να αξιολογήσει όλα τα κράτη αλλά και περαιτέρω διότι δεν είναι δυνατόν το εθνικό δίκαιο και τα εθνικά δικαιώματα τα οποία υφίστανται στα κράτη-μέλη να διαγραφούν. Αυτό δεν είναι δυνατόν να ισχύσει και μάλιστα ε, θα ήταν απλώς προς όφελος των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που θα θέλαν να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση για να κινούνται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ήθελα να σας πω προς το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όλα αυτά μας τα είπατε με μεγάλη σαφήνεια και μας εξήγησε για τη σχέση της δουλειάς μας με τη σχέση της νομικής επιτροπής. Πρέπει να ε, ε, βιαστούμε γιατί πλησιάζει η, η ώρα που θα έρθει ο Επίτροπος 10.30 θα πρέπει να μιλήσουν βέβαια και οι ε, εισηγητές, οι πέντε σκιώδεις εισηγητές αλλά προσοχή γιατί όσο πιο πολλοί μιλήσουν τόσο λιγότερο θα έχουν και οι άλλοι τρεις-τέσσερις συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τον λόγο Παρακαλώ να είστε συνοπτικοί. Και πρώτος θα ζητήσει το λόγο ο κύριος Ροσφόρ. Θα προσπαθήσω, συνάδελφε, να είμαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός και θα ήθελα να σας πω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την έρευνα του καθηγητού όπως είπατε έχουμε εδώ ένα συγκριτικό πίνακα για τις, για τις 19 19-22 ε, πάρα πολύ συνθετικά είναι εδώ τα πράγματα για να δούμε ε, ευθύς εξ αρχής τι μας απασχολεί και όπως τα είπε και η Ευλήν θέλουμε ελάχιστη ή μεγίστη εναρμόνιση. Όταν διαβάζουμε επομένως την έκθεση των δύο καθηγητών διαπιστώνουμε ότι η Wallis θέλει ελαχίστη και ο Σουάμπ μεγίστη εναρμόνιση. Εγώ βρίσκομαι στη μέση. Καμιά φορά είμαι πιο κοντά στην Wallis, αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι κάποιες ε, ρυθμίσεις θα πρέπει να παραμείνουν. Χρειάζεται όμω μία μεικτή λύση στην εναρμόνιση. Να υπάρχει μεγίστη εναρμόνιση εκεί όπου προκύπτει κάποιο πλεονέκτημα. Εκεί που κάνει καλό. Όπου εκεί μπορούμε να αναπτύξουν περισσότερο την αγορά χωρίς να συγκρίνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ προστασίας του καταναλωτή και δυναμισμού της οικονομίας. Ίσως τα πράγματα είναι απλούστερα στη δική μου χώρα, γιατί η Γαλλία έχει υψηλό επίπεδο προστασία καταναλωτού, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει δυναμισμό στην κατανάλωση. Μας κατηγορούν οι γείτονε ότι είμαστε πιο πολύ προσανατολισμένοι στην κατανάλωση και όχι στις άλλες μεταβλητές της οικονομικής ανάπτυξης. Όμως, εμείς νομίζω μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι έχουμε συγκεράσει την προστασία του καντών του με την δυναμική οικονομία. Και ταυτόχρονα έτσι τονώνεται η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές αυτά που έχουν ανάγκη, γιατί τα έχουν ανάγκη ασχέτως της ε, εμπιστοσύνης γιατί υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που έχει οριμάσει η κατανάλωση και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ακριβώς όπως ακούμε για τους νέους τομείς όπως η πληροφορική. Εκεί διαπιστώνουμε τι γίνεται, ότι οι καταναλωτές ε, κινούνται ανάλογα με την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην αγορά. Είπαμε για την απορρίθμιση της αγοράς, ε, ας πούμε για με το, το, το, το, ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, διότι έχουν δυσπιστεί προς τους διαφορετικούς operators οι καταναλωτές όταν επομένω δεν είναι τόσο σίγουρο για το τι γίνεται. Και γι' αυτό και έχουμε 96% των ε, ε, καταναλωτών οι οποίοι μένουν στη ΔΕΗ και δεν πάνε στους ε, εναλλακτικού operators. Οπότε έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, έχουμε 1600 συνολικά. Και εγώ έχω καμιά εκατοστή και να σας πω τα βασικά σημεία τώρα ότι την ε, Τρίτη θα άρχισει η δουλειά για να δούμε για το τέταρτο κεφάλαιο τι συμβαστικές τροπολογίες μπορούμε να έχουμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία. Δεν λέω ότι θα συμφωνήσουμε με όλα, αλλά πάντως πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, ε, για την προσπάθεια που κάνει, για τις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε κι άλλο. Ε, μας τα είπε και ο Ανδρέας ότι ακριβώς το 4 είναι το σημείο της ισορροπίας μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης ε, εναρμόνισης. Προσωπικά Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, να ε, περισσωθούν και πιστοί από τη μέγιστη αρμόνιση όπως για την παράδοση του αγαθού, αγαθού για τον ε, ε, για, τη μετακύληση του κινδύνου, κάποια τέτοια σημεία και ίσως το πιο στρατηγικό είναι το άρθρο 26 εκεί που αφορά τα ένδικα μέσα όσον αφορά κάποια ελαττώματα τα οποία προκύπτουν στη σύμβαση Οπότε να δούμε και σε ποια σημεία χρειάζεται στην αρμόνιση. Αυτά θα τα συζητήσουμε με τον εισηγητή. Κατά τη γνώμη μου πάντως ε, δεν θέλω να υπάρχει μια ιεράρχηση αυτών των ε, ενδίκων μέσων γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που υπάρχει ελεύθερο δικαίωμα του καταναλωτού να διαλέξει με ποιο μέσο θα αποζημιωθεί για το ελάττωμα το οποίο προέκυψε προσοχή, να μην το θέσουμε αυτό ένα αμφιβόλο, γιατί αυτό θα είναι ένα χτύπημα ε, στα δικαιώματα του καταναλωτή από την άλλη μεριά, ε, κάτι το οποίο προελέχθη για τα, άρθρα, για τα κεφάλαια 2 και 3 εγώ θεωρώ ότι όλα πάνε καλά και είναι πολιτικοί οι λόγοι γιατί προφορώ, προτιμώ αυτή η οδηγία να προχωρήσει ε, όσο μπορεί. Να προχωρήσει δηλαδή σε βάθο έστω και με περιορισμένο πεδίο εφαρμογή Από την άλλη μεριά, εάν συνενώσουμε το 2 και το 3, τότε θα έχουμε προχωρήσει όσον αφορά την πώληση εξ απόσταση και εδώ είναι το στοιχείο στο οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά και έτσι να έχουμε από την άλλη μεριά για τις προσυμβατικές πληροφορίες ε, λιγότερη πρόοδο και κυρίως όσον αφορά τις πωλήσει σε κάποιο εμπορικό χώρο, σε κάποιο κατάστημα έχοντας προχωρήσει στο στρατηγικό το θέμα εκείνο. Ακριβώς εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Και χρειάζεται να δούμε τι γίνεται και με τις νέες μορφές εμπορίου όπως οι πωλήσει εξ αποστάσεως. Όλα αυτά θα τα ξαναεξετάσουμε και είπαμε ότι ξεκινάμε με το κεφάλαιο 4 όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει με το δεξί γιατί έχουμε την πρώτη συμβαστική τροπολογία. Πρόεδρος, συμφωνώ μαζί σου. Κύριε Ρούλη. Δεν ήξερα ακριβώς το timing της συνεδρίας, δεν είμαι έτοιμο.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 από αυτό θα επηρεαστεί συγγνώμη, και η αγορά των ε, πολιτών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο. Ε, Βεβαίω υπάρχουν και πάρα πολλέ τροπολογίε. Ε, ε, αναρωτιέμαι αν μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουμε λίγο τον αριθμό αυτό και αν μπορούμε και να μειώσουμε ε, και τα σημεία τα οποία μας δυσκολεύουν περισσότερο στο κείμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσουμε όλα τα στοιχεία και ε, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δουλέψουμε ε, πολύ στις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών. Όσον αφορά τώρα την ε, μορφή ε, της ε, οδηγίας, τα κεφάλαια 2 και 3 μπορούν να συμπτυχθούν και επίσης το η αναφορά στις ε, γενικές ε, ε, προϋποθέσεις με έναν οριζόντιο τρόπο με βρίσκει σύμφωνο. Παρόλα αυτά φοβούμαι ότι ενδεχομένως κάποια στοιχεία θα χαθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει λόγος βεβαίως ε, για μεικτή εναρμόνιση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ε, θα πρέπει και η εργασία μας να είναι πρακτική και να είναι εύκολο να αναλυθεί. Ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τα θέματα της συμμόρφωσης και να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο βαθμό συνοχής και συμφωνίας εκεί που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε απολύτως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κύριο μέλημά είναι άλλωστε η προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Τα άρθρα 26 και 28 είναι τα πιο δύσκολα κατά την άποψή μου. στο άρθρο 26 δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αυτό θα σημαίνει ότι μειώνουμε την περαιτέρω φυστάμενα υφιστάμενα όρια και νομίζω ότι θα πρέπει ε, να γίνει εδώ αναφορά σε όλες τις δυνατότητες, δηλαδή είτε επιστροφής, είτε ε, αλλαγής, είτε και επιστροφής των χρημάτων για το άρθρο 28 που αναφέρεται ε, στην ευθύνη της ε, επιχείρησης ε, υπάρχει μια τροπολογία που έχουμε υποβάλει στο σημείο αυτό. Εμείς θέλουμε να επιμηκυνθεί η περίοδος από τα 2 στα 6 χρόνια. Κατά την άποψή μας 2 είναι πολύ λίγα υπάρχουν ε, μερικές φορές ε, ε, προϊόντα όπως ας πούμε τα κεραμίδια ή τα τούβλα τα οποία είναι, είναι δύσκολο να αξιολογηθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ελπίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκλείσουμε από την αγορά όλες αυτές τις εταιρείες ε, οι οποίες ε, τελικά προσφέρουν πολύ χαμηλής ποιότητος ε, προϊόντα. Επίσης όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται για την επιστροφή των προϊόντων νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια καθολική εξάμηνη περίοδο περίοδο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα, όλα όσα μας είπατε. Ούτως ή άλλως ε, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα δείτε με τον ε, εισηγητή. Δεν νομίζω πάντως ότι ο εισηγητής με ακούει αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία σημασία. <laughs> δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κύριε Σιγητά, μόλις χάσατε τις ε, παρατηρήσεις που σας έκανα. Ο κύριος Ρεδεφιλίδης. Το επιδιώκουμε βγαίνει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Επομένως θα περιοριστώ σε πέντε βασικές σκέψεις που διέπουν αυτές τις τροπολογίες. Ε, πρώτα θέλω να αναφερθώ στις ε, πληροφορίες για τα προϊόντα. Έχουμε την, επικεντρωθεί σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τιμών ε, είναι κρίσιμη σημασία ο καταναλωτής να γνωρίζει την τελική τιμή που θα καταβάλει συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Δεύτερον, για την περίοδο υπαναχώρησης. Βασική αρχή είναι η καθολική εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης με τις λιγότερες πιθανές εξαιρέσεις. Προτείνουμε επίσης την αύξηση της περίοδου υπαναχώρησης, ώστε αυτή να αντιστοιχεί με την περίοδο που έχει ο έμπορος για αντικατάσταση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του προϊόντος. Παράλληλα, εάν ο έμπορος δεν παρέχει σαφείς πληροφορίες στον καταναλωτή για το δικαίωμα επαναχώρησης, τότε αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί λόγω μη σαφούς προσδιορισμού και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαρκεί επαόριστο. Εδώ αξίζει να πούμε ότι η δυνατότητα επαναχώρησης κατοχυρώνεται ως δικαίωμα, άρα οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος βαραίνουν αυτόν που προσφέρει το δικαίωμα, δηλαδή τον έμπορο, και όχι αυτόν που απολαμβάνει το δικαίωμα. Τέλος, η έναξη της προθεσμίας θα πρέπει να ταυτίζεται χρονικά με τη χρονική στιγμή μεταφοράς του κινδύνου στον καταναλωτή. Τρίτον, σχετικά με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή για παραδείγμα αντικατάσταση, σε περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει το μέσο που τον συμφέρει άρα δεν θα πρέπει να επιτραπεί στον έμπορο η άρνηση αποκατάστασης. Αν αυτό συμβεί θα πρέπει να θεωρείται ως μη εκπλήρωση της σύμβασης. Ανάλογα και οι διατάξεις σχετικά με την παράδοση αποτελούν ευθύνη του εμπόρου, ώστε τα εμπορεύματα να είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, με εξαίρεση μόνο αν ο καταναλωτής συμφωνήσει εκ των προτέρων να λάβει αγαθά που δεν πληρούν τη σύμβαση. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει καθορισμός του τι ορίζεται έλλειψη συμμόρφωσης ελάσσονος σημασία ώστε να ξεκαθαριστεί πότε ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση του. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών, θα πρέπει να αρχίσει με ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή σε σταθερό εναπόθεμα. Οι ισχυρισμοί για έναρξη της παροχής υπηρεσίας αυτοβούλως από τον έμπορο δεν μπορεί να ισχύσει, μιας και δημιουργεί κενά ω προς την, προσπάθεια, προς την προθεσμία για την υπαναχώρηση από τον καταναλωτή. Κυριάκο, λένε οι διερμηνείς, εάν μπορείς να μιλάς πιο... Ναι, τελειώνω, τελειώνω, τελευταίο σημείο. Πολύ αργά θα στο το πω. Νομικές εγγυήσεις των δύο ετών, για μας αυτή η θέση είναι το κατόφλι και όχι η οροφή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρούν διατάξεις για εγγυήσεις τουλάχιστον δύο ετών. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Προσπάθησα να το πω γρήγορα για να ξεχνήσουμε χρόνο. Πάρα, πάρα πολύ εξέπαινο αυτό. Αλλά είναι και σημαντικό επίσης και να μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λες. Ωραία, τελειώσαμε τώρα με τους κοιόδες ηγητές και μας μένει ένα τεταρτάκι να ολοκληρώσουμε το θέμα για να μην φάμε το χρόνο του Επιτρόπου. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει το Συμβούλιο η Κομισιόν, η κυρία Ρότεβα, κύριο Σουάμπ, κυρία Σούλη, δεν θέλει κανεί άλλο να εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών και η κυρία Ντεγκρούπ και ο κύριος Κρότσμα. Παρακαλώ, δύο λεπτά ο καθένας. Δύο λεπτά, αλλιώς δεν γίνεται. Δύο λεπτά ο καθένας. Κυρία Ρόιτερ πρώτη. Πάρα πολύ θετικό είναι το ότι συμφωνούμε όσον αφορά την εναρμόνιση των πληροφοριών και μένα με προβληματίζει το θέμα του ψηφιακού περιεχομένου γιατί πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα υπάρχει διαφάνεια στις πληροφορίες για την διαλειτουργικότητα ε, των ηλεκτρονικών αγαθών ούτως ώστε να μπορεί να γνωρίσει κανείς κατά πόσον το software, το λογισμικό θα μπορεί να ε, είναι συμβατό με, τα, με Windows, τις διάφορες μορφές το Windows, τα XP κλπ. Τώρα, το άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι η μετακύληση της ευθύνης όσον αφορά την ανταλλαγή, όσον αφορά τα ανταλλακτικά, όσον αφορά τα διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν και όχι μόνο για τον καταναλωτή αλλά και για τους κατασκευαστάς, για ε, τα παιχνίδια και για άλλα προϊόντα. Τώρα, όσον αφορά τα εμπορεύματα, θα πρέπει να οριστεί το τι είναι ψηφιακό αγαθό και αυτό να γίνει ξεκάθαρα ε, σε σχέση επίση με τα αγαθά ή τα εμπορεύματα τα οποία τα κατεβάζει κανεί από το Ιντερνετ. Τώρα, κάποια κάποια προϊόντα δεν θα πρέπει να καλυφθούν, θα πρέπει να εξελιχθούν. τώρα δεν έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο. Ε, έχω 60 τροπολογίες κατεβάσει. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να εισηγητήσω τον... να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του και του εύχομαι καλή τύχη. Ah, suis Monsieur Κύριε Πρόεδρε, λέει συνολικά. αν ο κόσμος ήταν τέλειος θα χρειαζόταν μεγή στην αρμόνιση για τα πάντα. Γιατί αυτό θα έκανε ευκολότερη τη λειτουργία της ιστορικής αγοράς και έτσι θα είχαμε το τέλειο επίπεδο προστασίας του καταναλωτού ε, το, το καλύτερο δυνατόν ακριβώς ε, και θα υιοθετούσαμε το, το, το, το επίπεδο προστασία όπου υπάρχει τέλειο. Όμω δεν γίνεται αυτό, δεν είναι τέλειο ο κόσμο, άρα πάμε ε, αλλού μήνυμο, αλλού maximum ε, εναρμόνιση ε, για τα 5, 10 και 20 χρόνια τα επόμενα επομένως θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη ε, εκεί που, που ισχύει η ελαχίστη εναρμόνιση να αλλάξουν τα, τα, τα δικαιώματα και να θέσουν κάποιο στόχο, τόσο ώστε σε κάποια χρόνια να προχωρήσουν από την ελαχίστη στην μεγίστη εναρμόνιση και τότε να καθορίζεται το τέλειο επίπεδο προστασία του Έχω τρει παρατηρήσει για όλε αυτέ τι 1600 τροπολογίε. Ε, το, το, το, το, καλό ποτέ δεν βλάφτει, λέμε στη Γαλλία. Αλλά όταν όμως το, παρακάνουμε παραμπερδεύουμε την ε, κουβέντα οπότε πάρα πολύ σωστά τα, το, το θαυμάζω τον κύριο Σφάβ και όσον αφορά τώρα την υπαναχώρηση και τις σχετικές προθεσμίες νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την λευκή περίοδο όσον αφορά τις συμβάσεις οι, οι οποίες έχουν ε, συναυθεί ως συμβάσεις ε, από το σπίτι γιατί το θέμα το κρίσιμο είναι κατά πόσο κανείς είχε το διάστημα του, του να σκεφτεί και να αποφασίσει. Ε, επίσης όσον αφορά την ιεράρχηση αυτή όπως αναφέρθηκε ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για το 12 για το 92 ε, την τροπολογία 92 του κύριου Σφάμπ για να μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και επίσης κατά τρίτον ε, υπάρχει μια μικρή σύγχυση, είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα το ότι σε, υπάρχει κάποια ολόκληρη κατηγορία βιοτεχνών οι οποίοι ε, επί παραγγελία κατασκευάζουν κάποια κάποια, μπορεί να το είναι ένας επιπλοποιός, φτιάχνει ένα τραπέζι, μια καρέκλα, το κάνει με τα χέρια του μόνος του και του παίρνει δύο, τρεις, πέντε μήνες ε, δεν ξέρω, εάν λοιπόν για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και τη λειτουργία της αγοράς. Να μην έχουμε προβλήματα με, με, με, με κάποιες διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τη μαζική παραγωγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτος, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Κύριος Φαντεκάμπ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και οι οδησηγητές και ο κύριος Σουάμπ έχουν ε, καθορίσει το πού θα κινηθούμε. Δεν έχουμε χρόνο, επομένω να μείνουμε γρήγορα, αλλά θα ήθελα να σα ε, επισύρω την προσοχή στο, στην τροπολογία 13 αλλά και στην 24 και την υπαριθμόν 62 όσον αφορά την, ε, τα, τα θέματα μεγίστης και της αναμονήσεως όπως ε, προαναφέρθηκε και η κυρία Γκέμπχαρτ ετώνησε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών γιατί δεν μπορούμε να αδρανίσουμε ενώπιον αυτής της πρόκλησης αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Εκεί που μπορούμε να έχουμε μεγίστη εναρμόνιση, να το κάνουμε, να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα το 13 και το 24, το 1324 αφορά κάποια διαρκή αγαθά. Έπιπλα, εξοπλισμό οικιακό, και, και στο 1362 επίσης αναφέρεται η ανάγκη της μεγίστης ε, εναρμόνισης και η σχετική προθεσμία του 1,5 έτους. Μπράβο σας, είσαστε παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά το ότι το χρονικό όριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα και εγώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Αντρέα και για την εργασία του και για την ε, δυνατότητα προσαρμογής που διαπιστώσαμε, αλλά και την ε, πρόθεση να ακούσει προσεκτικά αυτά που του λένε οι άλλοι. Ε, Βεβαίω, εμεί έχουμε υποβάλει τροπολογίε υπέρ τη προστασία των καταναλωτών, κυρίω δε τη δυνατότητα επιλογή ε, του τρόπου επικοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα θέλουν επικοινωνία σε χαρτί ε, και είναι δικαίωμά τους. Επίσης θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία ε, μεταξύ του καταναλωτού και του, του αγοραστού τέλο πάντων και του κατασκευαστού ή πολιτού ε, όσον αφορά τα πολύ μικρά αντικείμενα. Όσον αφορά τώρα τη διασυνοριακή εμπορία νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ε, βαρύνουμε ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες κυρίως ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή να μην ε, υποχρεώνουμε τους πάντες να δώσουν, ακόμα και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να δώσουν κάποιες εκ των προτέρων πληροφορίες, οι οποίες θα βαρύνουν πάρα πολύ τη δουλειά τους Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να ε, ε, πετύχουμε μία προενεργητική ε, τάση του καταναλωτή. Ούτως ή άλλως ο καταναλωτής θα πρέπει πάντα να έχει την δυνατότητα να καταναλώσει ή να μην καταναλώσει. Είναι δικιά του απόφαση. Και επίσης, όσον αφορά το παράδειγμα της κυρίας Γκέπχαρτ, η οποία μας διηγήθηκε τα χρήματα τα οποία πληρώσανε, ε, πρώτον, να σημειώσω ότι ε, πολύ συχνά οι άντρε δεν προσέχουν αυτό το επιπλέον ποσό. Οι γυναίκε είναι πιο προσεκτικέ σε αυτή την περίπτωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, στη Γαλλία έχουμε το λεγόμενο διπλό κλικ. Δηλαδή, αν σα ζητήσουν διπλό κλικάρισμα για να αγοράσετε κάτι, να είσαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δίνετε τη συνένεσή σα και για κάτι άλλο. Δηλαδή, για να σα κρατήσουν περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια τη χρηματική συναλλαγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ε, ναι, αυτό το διπλό κλικ νομίζω ότι είναι μια καλή ε, αναφορά. Κύριε Λεγουίκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ γρήγορα ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας ε, κύριο Σφάμπα για τις άοπνες προσπάθειές του κατά τη διάρκεια των προηγουμένων εβδομάδων και ε, η εργασία του είναι πραγματικά αξιέπαινη και αξιοθαύμαστη γιατί ήταν πάντα στη διάθεση όλων, ήταν υπομονετικός, ε, μηχανεύτηκε πράγματα και πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έκανε πολύ σκληρή εργασία υπέρ της ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών που επιτρέπει βεβαίω την περαιτέρω αύξηση του οικονομικού δυναμικού της εσωτερικής μας αγοράς. Γιατί αυτό είναι ε, το, το διτό ας πούμε θέμα, ο διτός στόχος. Καλύτερη προστασία, καλύτερο επίπεδο προστασία των καταναλωτών αλλά και ανάπτυξη του δυναμικού, του αναπτυξιακού λέω δυναμικού των ε, δυνάμεων της ε, αγοράς. Ε, σήμερα θα ήθελα να εκφραστώ και εξ ονόματος του συναδέλφου Νταβιέναβα που πολύ ασχολήθηκε με το κείμενο αυτό και που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα και ζητά συγγνώμη γι' αυτό. Λυπάται λοιπόν για αυτή την απουσία, ε, αλλά θέλω να επιβεβαιώσω ότι σε τροπολογίες τις οποίες έχουμε ε, υποβάλει. Δεν θα αναφερθώ ξανά στα σημεία που ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι ε, και επί του οποίου συνενούμε και συμφωνούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας σαν γαλλική αντιπροσωπεία να έχουμε εξαίρεση ε, εξαίρεση όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός καταστήματος. Επίσης είναι σημαντικό ε, να ε, προβλεφθεί γραπτή δήλωση και όχι τηλεφωνική συμφωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας γιατί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα για κάποιους καταναλωτές οι οποίοι ε, ε, αισθάνονται λίγο παγιδευμένοι εάν συμφωνήσουν για μια αγορά που τους έχει προταθεί από το τηλέφωνο. Επίσης, άρθρο 3 που επιτρέπει στις, θέλουμε να επιτρέπει στις χώρες μετά από πληροφόρηση και της Επιτροπής και των άλλων χωρών να λάβουν συγκεκριμένα περαιτέρω μέτρα για ε, πολύ συγκεκριμένα ε, σημεία αναθεώρησης του κειμένου. Ε, κατά την άποψή μας, με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε και τις μάλλον ηρεμούμε, καθησυχάζουμε ε, και τις, ε, τους καταναλωτές ε, και τους οργανώσεις των καταναλωτών, αλλά και καθησυχάζουμε τις ανησυχίες των υπολείπων κρατών μελών. Uh, Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ουσιαστική ερώτηση σε όλους τους ομιλητές. Ξεκινώ από αυτό που είπε ε, η κυρία Γκέπχαρ, ότι θέλουμε μία οδηγία προστασία των καταναλωτών. Πώς θα βοηθηθεί ο καταναλωτών όταν θα κάνει συναλλαγές εξ αποστάσεως. Οπότε θα έπρεπε τότε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση, γιατί σε όλες τις συζητήσεις για την εσωτερική βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές χώρες οι οποίες πλήττονται. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία πρόοδος για τους καταναλωτές, για την εσωτερική αγορά αλλά και για τους κατασκευαστές, διότι οι, έμποροι δεν παραδίδουν αν δεν είναι και αυτοί ασφαλείς. Διαφορετικά όλα τα άλλα τα οποία δημιουργούμε είναι απλώς γραφειοκρατία. Ε, θα πρέπει σαν ε, καταναλωτής να πάσα στιγμή να κοιτώ τι ισχύει για μένα. Γι' αυτό και ε, δεν συμφωνώ με τις πωλήσει πόρτα-πόρτα μέσω πλασχέδι διότι είναι κάτι τελείως εσωτερικό και κάθε φορά φορά που ε, συζητάμε εκεί για εναρμόνιση μας ε, λέγουν ότι πρέπει να ρωτήσουμε τις επιχειρήσεις αν το δέχονται ή όχι. Άρα πιστεύω ότι το δικαίωμα του καταναρωτή στην εσωτερική αγορά είναι να προστατεύεται εφόσον πληρώνει αυτός ο οποίος καταναλώνει. Δεν πρέπει λοιπόν ε, να πάνε οι απαιτήσει πάρα πολύ ψηλά διότι τότε θα ε, ε, έχουν αντίκτυπο στις τιμές των προϊόντων. Θα ήθελα να σκεφτείτε αυτά τα σχόλια όταν μιλάτε για εναρμόνιση στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Η κυρία Κοράτσα, ο κύριος Μάντερς αλλά ο κύριος Σταγιάννη αργεί λιγάκι και έτσι μπορώ να δώσω στην κυρία Κοράτσα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες αλλά η προστασία των καταναλωτών δεν συνεπάγεται προστατευσισμό. Αυτό είναι απειλή για τους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε το όραμά μας του δημοσίου συμφέροντας και αυτό είναι η εναρμόνιση. Όπως είπε και ο κύριος Ροσφόρ, ο δυναμισμός οικονομικά συνάδει ε, με την προστασία των καταναλωτών διότι ο κατακαιρματισμός είναι κατά των ε, καταναλωτών δεν πρέπει να προσιλωθούμε μόνο σε θέματα ε, ιδεολογιών πρέπει να στηρίξουμε τον εισηγητή ο οποίος αποβλέπει σε μια ρεαλιστική ρεαλιστική συνενετική λύση και θα ήθελα να προειδοποιήσω τους συναδέλφους τι θα συμβεί εάν αποδυναμώσουμε αυτή την οδηγία. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους λαούς της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη απειλή είναι ο προστατευσισμός και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια κατάσταση η οποία να είναι προς όφελος και των επιχείρησεων αλλά και των καταναλωτών. Ευχαριστώ και ο κύριος Μάντερς τέλος. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας θυμίσω την ε, συμβουλή του κυρίου Μόντι σελίδα 92 ότι θα έπρεπε να ρυθμίσουμε διάφορα θέματα περίπλοκα και ελπίζω θα επιτύχουμε και εδώ και δεύτερον, συμφωνώ με τον κύριο Βαντεν Καμπ ότι πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Και τέλος, εύχομαι στον Ανδρέα Σβάμπ καλή επιτυχία για να μπορέσει να υπάρξει συμβασική λύση σε τόσο πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα είναι καταρχάς θα έπρεπε να έχω χαιρετήσει πολύ πιο πριν το Συμβούλιο. Τώρα ήρθε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε ε, χρήσιμο θα ήταν να ζητήσουμε από τον κύριο Άντενχοφ ο οποίος ε, είναι επικεφαλής της υπεύθυνη ομάδος να μας πει πού βρισκόμαστε και μετά ε, θα επανέλθω μετά από, το, τα διάφορα σχόλια στον εισηγητή για να καταλήξει. Ε, θα βάλω το ρολόι μπροστά εάν ε, μου επιτρέπετε για να σας υπενθυμίσω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Είναι σαφές ε, στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να εργαστεί σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ε, έχω διαβάσει όλες τις τροπολογίες, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε τι κάνει το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και την ε, θέση ε, και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην ε, συζήτηση. Μέχρι τώρα είχαμε 15 συναντήσεις της ομάδας εργασίας και πολλές συζητήσεις. Βεβαίως θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση, να ξέρουμε ποια είναι η άποψη όλων, έχοντας ακούσει ε, εκτάσει της απόψεις ε, όλων των συμμετεχόντων στον ε, διάλογο. Εάν τα καταφέρουμε θα είναι εξαιρετικό. Βλέπουμε με μεγάλη προσοχή και παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν στο Κοινοβούλιο και τι γίνεται και στα κράτη-μέλη, γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε την οδό της συνένεσης. Ελπίζω ότι τη 10η Δεκεμβρίου θα υπάρξει συμφωνία. Άκουσα ότι ε, τα πράγματα μάλλον ε, θα προχωρήσουν ε, καλά και μην ξεχνάμε ότι ειδικά για θέματα προστασίας καταναλωτών οτιδήποτε επιπλέον θεσπιστεί είναι καλό τα κεφάλαια είναι ισορροπημένα και πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ελπίζω ότι 10 Δεκεμβρίου να μην έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ και ξέρω ότι δουλεύετε πολύ και με τους εισηγητές και γνωρίζετε πολύ καλά το τι συμβαίνει. Ε, θα συζητήσουμε το θέμα με τους ε, συντονιστές βέβαια και όπως μας είπατε θα συναντηθείτε την 10η ε, Δεκεμβρίου ενδεχομένως δε ο αρμόδιος υπουργός να είναι και στην Ολομέλεια παρών εκπροσωπώντας την Προεδρία, κάτι τέτοιο άκουσα και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Um, now, ο κύριος Πέτρη, σε δύο λεπτά αν είναι δυνατόν. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. We uh, Όντω, πρόκειται εδώ πέρα για μια μεγάλη πρόκληση. Το πώ η Επιτροπή σα και, και ο εισηγητή συγκεκριμένα θα μπορέσει να το καταφέρει με όλε αυτέ τι ε, τροπολογίε που πάνε προ όλε τι κατευθύνσει και με τη σειρά μου ε, θα πρέπει και εγώ να σας πω ότι συμφωνώ σε αυτά που είπε η κυρία Κράτς ε, ε, και ο κύριος Ροσφόρς για το ότι δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνά κανείς την προστιθεμένη αξία της πλήρους εναρμόνισης βεβαίως και υπάρχει χρησιμότητα σε στην εναρμόνιση και προσπαθεί προς αυτήν την κατεύθυνση ο εισηγητής για το πώς θα έχουμε την εναρμόνιση, πώς θα έχουμε την ε, καλύτερη προστασία του καταναλωτή σε σχέση με την πρώτη μας ε, πρόταση να δούμε πώς θα έχουμε ε, ευχαριστημένους και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις Ελπίζω ότι στις διαπραγματεύσεις θα τα βρούμε. Τώρα όσον αφορά τα επιμέρους κεφάλαια, ε, συμφωνούμε εμείς με αυτούς που θέλουν την πλήρη εναρμόνιση για το κεφάλαιο 3 και βεβαίως ε, αναγνωρίζουμε το ότι υπάρχουν κάποια σημεία του κεφαλαίου 4 όπου θα πρέπει να διερευνηθεί ακόμα το τι θα κάνουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την μετακύλυνση του κινδύνου σε σχέση με το πόση εναρμόνιση θα κάνουμε επίσης θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι ανέκαθεν το Κοινοβούλιο σχέση με το Συμβούλιο είναι πρωτοπόρο όσον αφορά την εναρμόνιση. Ε, να μην το ξεχνούμε αυτό. Το Συμβούλιο πάντως ε, βρίσκεται στη σωστή ρότα και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να ξεχνά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, να μην ξεχνά ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση. Ο Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα, κύριε Σουάμπ, τι θα θέλετε να μας εξηγήσετε με συντομία. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει έτσι σοβαρή συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι πολλά ενδιαφέροντα σχόλια έγιναν και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να καλύψουμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων, μεσαίων μεγέθους επιχειρήσεων και ε, γι' αυτό ο, πολλοί θα μπορούν να υποφεληθούν Δεύτερον, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ρομπέρο Φορ. Δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ καλής προστασίας των καταναλωτών και υψηλού βαθμού ασφαλείας. Άρα θα προσπαθήσω να βελτιώσω τα κεφάλαια 2 και 3. Προσλέπω και στι περαιτέρω συζήτηση και όσον αφορά τα ψηφιακά προϊόντα που ανάφερε η κυρία Γκέπχαρτ και Ρόιτοβα ήθελα να κάνουμε μία ακρόαση δεν τα καταφέραμε αλλά είναι ένα πολύ περίπλοκο ε, νομικό και ουσιαστικό θέμα και δεν ξέρω αν εκεί θα επιτύχουμε αλλά προσβλέπω σε όλες τις συζητήσεις και είμαι ευγνώμων για οποιοδήποτε σχόλιο και έστω και οποιαδήποτε κριτική. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο θέμα αυτό. Ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο και ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι ε, προχωρήσαμε καλά και η πρόοδος μας είναι ικανοποιητική. Ε, βλέπω εδώ το, την εκτελεστική περίληψη αυτής της εκθέσεως που είναι χρήσιμη. Όταν λοιπόν κοιτούμε ε, και προσβλέπουμε στην εναρμόνιση προσπαθούμε να βρούμε τους τομείς όπου θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το διασυνοριακό εμπόριο χωρίς να μειώσουμε την προστασία του καταναλωτή όλα αυτά είναι θετικά και είναι ένα καλό σημείο κινήσεως για τον εισηγητή και καλό θα ήταν να έχουμε συμφωνία στα σημεία 2 και 3 διότι όπως είπατε κύριε εισηγητά αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι θα πρέπει ε, να εστιαστούμε ε, τα, στις διασυνοριακές συμβάσεις πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε σήμερα αλλά θα δούμε πού θα καταλήξουν οι συμβιβασμοί. Κατόπιν των συζητήσεων θα ήθελα και εγώ να γνωρίζω πού μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι για να να υπάρχει ανώτατη εναρμόνιση ή ακόμη και ελάχιστη εναρμόνιση διότι εδώ μιλάμε για την προστασία του καταναλωτή και προσπαθούμε να δώσουμε ίσους καταναλωτές ε, την ελάχιστη ε, προστασία την οποία δικαιούνται και ε, συμπεριλαμβανομένης ε, και, και, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συνδυάσουμε και προστασία των καταναλωτών και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε σε όλους τους κοιόδης εισηγητές και τον ε, ουσιαστικό κύριο εισηγητή ε, καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Προχωράμε τώρα εις ε, την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κύριο Ταγιάννη. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ σήμερα για να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα εργασίας σας για το 2010-2011 και τις αρμοδιότητές σας ε, που είναι ε, ουσιαστικά η βιομηχανία και η επιχειρηματικότητα ε, σχετικά να μας μιλήσετε για τα βιομηχανική στρατηγική είδαμε ότι έχετε προχωρήσει πολύ καλά ακούσαμε πολλές προτάσεις όσον αφορά ιδίως τα αυτοκίνητα οχήματα ε, και ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε και άλλα προγράμματά σας. Σας ευχαριστώ. Εχθές το βράδυ ήσασταν υπεύθυνο ε, για ένα πολύ σημαντικό γεγονός αλλά σήμερα το πρωί που ήσασταν εδώ μαζί μας δεν θέλαμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήμουνα πολλά χρόνια μέλος του Κοινοβουλίου και πράγματι χαίρομαι κάθε φορά που ε, έρχομαι, ε, κάθε φορά που έρχομαι εγώ εδώ χαίρομαι πάρα πολύ. French cuisine and Mediterranean ε, βεβαίως ξέρετε εδώ είμαστε και πολύ ε, μεσόγειοι, εγώ ασχολούμαι και με τη μαγειρική, μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα από την ιστορία μας, και θεωρώ ότι όλη αυτή η κληρονομιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε, εγώ μιλάω συνήθως τη γλώσσα μου και αυτό θα κάνω και τώρα. Και μια και υπάρχει διερμηνία, μπορώ να το κάνω άνετα. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό, όπως θυμήσατε και εσείς, στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ενδιαφέρον, λέω, να έχω την δυνατότητα να σας μιλήσω για το πρόγραμμα εργασίας του επόμενου έτους. Η διεθνής οικονομική κρίση που έπληξε την Ευρώπη και μάλιστα σε βάθος, οπωσδήποτε συνέλαβε, συνέβαλε συγγνώμη, στην τροποποίηση των προτεραιοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 και ε, βεβαίως οι οικονομικές προκλήσεις και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο σύνολό τους πλέον έχουν μια πάρα πολύ σημαντική θέση στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα έτη μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σε αυτή τη νέα στρατηγική η οικονομική ανταγωνιστικότητα δεν αφορά μονάχα συγκεκριμένο και διαρκές μέλημα, αλλά αφορά πλέον μια πολιτική προτεραιότητα και με την εφαρμογή των εμβληματικών πρωτοβουλειών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα παρουσίασε όσον αφορά την ε, εσωτερική αγορά, την καινοτομία και την βιομηχανική πολιτική, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξαναφέρει την, Επιτροπή, συγγνώμη, την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στην οδό της ανταγωνιστικότητας. βιομηχανική πολιτική. Το έγγραφο το οποίο ενεκρίθη την 28η ε, Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους ε, λαμβάνει υπόψη τις ε, κύριες τροποποιήσεις που επηρέασαν την παγκόσμια οικονομία και επομένως και την ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς εστιάσαμε ξανά την προσοχή μας στην βιομηχανία και στην επιχείρηση ως μέσο και εργαλείο ανάπτυξης δημιουργίας θέσεων εργασίας μετά από πάρα πολλά χρόνια κατά τα οποία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, και οι υπηρεσίες αποτέλεσαν κέντρο ε, όλων των προσπαθειών ανάπτυξης και ε, είδαμε βεβαίως που μας οδήγησε αυτό ξέρουμε πλέον ότι όχι ότι βεβαίως δεν θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο οι υπηρεσίες ή οι τράπεζες αλλά ότι θα πρέπει και άλλοι τομείς να συνεισφέρουν στην πραγματική οικονομία και άλλωστε αυτό αναφέρεται και στην συνθήκη της Λισαβόνας ότι θέλουμε μια αγορά η οποία θα έχει στόχο την κοινωνική πολιτική και επομένως θα πρέπει ε, να εργαστούμε και το θύμισε άλλωστε και ο κύριος Σφάμπ πριν από λίγο πρέπει να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε μαζί ε, με, ε, με καλύτερο ανταγωνισμό, λιγότερη μόλυνση, καλύτερο περιβάλλον να υπάρξει και ένας πολύ σημαντικός πρωταγωνιστικός χώρος και ρόλος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να δοθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων που θα πρέπει ε, να έχει η ε, βιομηχανία. Ε, στη νέα προσέγγιση εμείς δεν θέλουμε απλώς να λάβουμε υπόψη κάποιες εθνικές αλυσίδες αξιών, αλλά θέλουμε ολοκληρωμένη διαδικασία από τις πρώτες ύλες μέχρι την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και ε, βεβαίως η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον πραγματικότητα και επομένως θα πρέπει να δούμε πέρα από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει όταν μιλάμε για αγορά να αναφερόμαστε στην παγκοσμιοποιημένη αγορά ε, και βεβαίως θα αναφερθώ στην εσωτερική αγορά αργότερα. Ε, θα ξεκινήσουμε μέσα από τις δράσεις για την τυποποίηση και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουμε και νέες αγορές. Έλεγα λοιπόν ότι απέναντι στην ε, παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι ε, και επομένως χρειάζεται όλο και περισσότερο μια, ένας συντονισμός όσον αφορά ε, τις πολιτικές ε, και βεβαίως είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βάσει και της αρχής επικουρικότητας και οι αρχές ε, των κρατών μελών. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να συντονίσει και να κάνει πιο ανταγωνιστικό και λειτουργικό το όποιο σύστημα. Ε, στην ανακοίνωση έχουν ε, ε, αναφερθεί πολλά εργαλεία, πολλά μέσα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που μόλις ανέφερα. Μιλάμε για ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς, μιλάμε για βεβαίως αναθεώρηση της τυποποίησης, τεστ τα οποία θα είναι τεστ ανταγωνιστικότητας, τα οποία θα είναι πιο ανταγωνιστικά και τα οποία θα είναι ενισχυμένα γιατί θα έχουν πλέον αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα ε, αφορούν τι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει ε, και τη ενίσχυση της κυβέρνηση, έτσι όπω αυτή αναφέρεται στο άρθρο 173 της Συνθήκης Λισαβόνα. Ε, εσωτερική αγορά είναι βεβαίω ένα θέμα το οποίο αφορά όλου μα και το οποίο κυριότερα αφορά την Επιτροπή σα εδώ. Όλοι θέλουμε μια πιο δυνατή εσωτερική αγορά και πιο εμβαθυμένη εσωτερική αγορά γιατί αυτό είναι κάτι ουσιώδες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου μου Μισελ Μπαρνιέ ενέκρινε το Single Market Act, νέα πράξη, συγγνώμη, ε, ε, πράξη για την νέα αγορά. Μια σειρά δηλαδή από οριζόντιες πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν όλους τους τομείς ε, αρμοδιότητας των διαφόρων επιτρόπων και στόχο έχουν να καλύψουν τα χάσματα της εσωτερικής αγοράς. Εγώ πέρα από αυτά που ανέφερε ήδη ξέρω σε εσά στα πλαίσια μιας ακρόασης ο συνάδελφος Μπαρνιέ θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα οποία αποτελούν δικιά μου ευθύνη. Πρώτα απ' όλα η εποπτεία της αγοράς προϊόντων. Πρώτα απ' όλα και όσον αφορά την, τη δικιά μου αρμοδιότητα. Εγώ ε, δεσμεύομαι να σας ε, αναφέρω ε, διαρκώς και να σας ενημερώνω για όλες τις πρόοδους που έχουν γίνει όσον αφορά τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και που βεβαίως στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή αλλά και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών μας. Θέλουμε στην ουσία δηλαδή ασφαλή προϊόντα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι δέσμοι τιμή των, ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων που αναφέρεται και ως νέο κανονιστικό πλαίσιο, New Legislative Framework, ε, ε, ολοκληρώνει ε, και τελειοποιεί την, ε, το νομοθετικό κοινοτικό πλαίσιο όσον αφορά ε, την εποπτεία και την διεμπόρευση των βιομηχανικών προϊόντων. Είναι ένας νέος κανονισμός επίσης που αφορά το, την δέσμη που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010 και βεβαίως ο έλεγχος και η εποπτεία δεν αφορά μονάχα τη δικιά μας αγορά και τα προϊόντα τα οποία γίνονται στη δικιά μας αγορά αλλά και αυτά τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, κυρίως αναφέρομαι ε, στα μηχανήματα και τα ε, ε, παιχνίδια. Κατά αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μία δέσμη από προτάσεις 10 οδηγιών βάσει της οποίας που θα ευθυγραμμίζουν με την απόφαση 768 του 2008 και που θα καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο διεμπόρευσης και βεβαίως θα αφορά και διάφορους στόχους και διάφορους τομείς όπως η ηλεκτρονική, τα μηχανήματα σε εργαλεία μέτρησης, εκρηκτικά για μη στρατιωτικού σκοπούς, πυροτεχνήματα και άλλα συναφή, καθώ και ανελκυστήρε. Ε, βεβαίως γνωρίζομαι ότι ε, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όλες, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν έτσι ώστε να έχουμε ένα σύστημα συνεκτικό, ένα σύστημα ισόρροπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να περιοριστούμε μονάχα σε κάποιε σποραδικέ και στοχευμένε πράξει, Θα πρέπει να κάνουμε μια συνολική δράση. Γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός πολιετούς προγράμματος εποπτείας της αγοράς που θα επιτρέπει την ταυτοποίηση δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν μακροπρόθεσμα ε, και που βεβαίω θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του κατάλληλα χρηματικά ε, ποσά, κατάλληλους χρηματικούς ε, πόρους έτσι ώστε να διασφαλίσει έναν ικανό βαθμό αυστηρότητας των ελέγχων που θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη και συμβατή σε όλες τι χώρε μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διασφαλίσει στους ε, ε, οικονομικούς ε, φορείς ένα σωστό ανταγωνισμό, να μειώσει την απάτη και την παραχάραξη, την απομίμηση, να διασφαλίσει, να εγγυηθεί την σωστή και ενιαία αγορά των κοινοτικών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, RAPEX. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τιτάνιο έργο έτσι ώστε να μπορέσει προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί καλύτερα. Κατά αυτήν την ε, έννοια θα ήθελα ε, να ε, πω ότι μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα κυρίως των πιο ευάλωτων καταναλωτών, δηλαδή των παιδιών. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μέσω της νέας οδηγίας να αποκλείσει την χρήση επικίνδυνων ουσιών. Αναφερόμαστε λοιπόν σε όλες τις ουσίες οι οποίες είναι καρκυρογόνες, μεταλλαξιογόνες και επικίνδυνες για την ε, αναπαραγωγή καθώς επίσης και την κατάρκηση όλων των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών και των βαρέων μετάλλων. Ε, το έχω ξαναπεί ε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στην ακρόαση που είχαμε εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ότι δηλαδή θα πρέπει να ε, έχουμε μια διαρκή προσαρμογή ε, της, ε, των κανονισμών και των νόμων βάσει των νέων επιστημονικών στοιχείων που μας δίνονται έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Και αναφέρομαι εδώ ας πούμε σε την κατάργηση χρήσης υλών όπως το κάτμιο ή το ομόλυβος, ας πούμε. Ε, αλλά βεβαίως όσο και αν είναι αυστηρή ε, η νομοθεσία τίποτα δεν θα κάνει αν δεν εφαρμοστεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένο ότι και τα κράτη-μέλη έχουν ουσιοδέστατο ρόλο ε, να παίξουν κατά αυτή την έννοια. Όπως έχω ήδη πει επανειλημμένα, εγώ άοκ να προσπαθώ να συνεχίσω τις προσπάθειες αυτές έτσι ώστε να διατηρήσω την πίεση για να επιτύχουμε τον προκαθορισμένο στόχο μας, δηλαδή ε, ένα, υψηλό επίπεδο προστασίας ε, για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη και διαφάνεια ε, για τους εμπορευόμενους. Είμαι ευτυχής που και το Κοινοβούλιο κατανοεί αυτήν την κατάσταση και έχει ξεκινήσει μια σειρά μελετών και οργανώνει βεβαίως και συναντήσεις έτσι ώστε να εξελιχθούν σωστά τα πράγματα κατά αυτήν την έννοια. Το σήμα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, μέσα στα πλαίσια των προλεγωμένων μου είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό και παίζει σημαντικό ρόλο για την σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Μετά από ρητό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια εκστρατεία πληροφόρησης για το σήμα CE που αφορά ε, τους, όλους τους οικονομικούς φορείς, κυρίως δε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές. Και τον προηγούμενο Απρίλιο ε, σας ε, είχα πληροφορήσει ότι έχει ξεκινήσει η εκστρατεία αυτή, η οποία θα λάβει χώρα το 2010 και το 2011. Η ανάλυση μας καταδεικνύει ότι μπορεί κανείς να επιτύχει μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων, ενισχύοντας το ήδη ισχύον καθεστώς του σήματος ε, e, ε, και με άλλους τύπους ε, ελέγχου προϊόντων, ας πούμε έλεγχο στα σύνορα ή εποπτεία της αγοράς. Επαναλαμβάνω ότι βεβαίω εμείς σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις όσον αφορά το σήμα CE και όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της τυποποίησης. Επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το ε, θέμα αυτό και μάλιστα και στην ακρόαση που είχατε οργανώσει τον προηγούμενο Ιούνιο. Εν τω μεταξύ το Κοινοβούλιο ε, δείχνοντας μεγάλη πολιτική ευφυΐα εξέφρασε σαφώς την θέση του με την έκθεση πρωτοβουλίας ε, Κοζούκνιτς που πρόλαβε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση αντιπροσωπεύει σημαντική συμβολή στην εργασία αξιολόγησης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση της ε, τυποποίησης που όπως γνωρίζετε ε, θα ε, περιλαμβάνει και τον τομέα των ΤΙΚ και που προτιθέμεθα να εγκρίνουμε περί τον Απρίλιο του 2011, τον επόμενο Απρίλιο δηλαδή, μία δέσμη η οποία θα, αφορά, θα περιλαμβάνει ανακοίνωση και κανονισμό και ε, που ε, θα βάλει σε ένα ε, νομοθετικό μέσο τις, τα τρία παρόντα μέτρα. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο σύστημα τυποποίησης, ένα δυναμικό σύστημα τυποποίησης που θα έχει ε, την δυνατότητα και να ε, διασφαλίσει την διαλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και να συμβάλλει στην καινοτομία. Ε, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξάγουμε την, τα τυποποιημένα μας προϊόντα και με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις μας θα είναι σε θέση να ανοιχνεύσουν καλύτερα τις αγορές πέραν της εσωτερικής αγοράς και βεβαίως και στα πλαίσια του διαλόγου ε, που υπάρχει και με την ε, Ρωσία πρέπει να σας πω ότι ήρθα σε επαφή με τον Υπουργό βιομηχανίας της χώρας αυτής ε, και ε, πρέπει να σας πω ότι στη χώρα αυτή από το 25% της έγκρισης των ε, ευρωπαϊκών στάνταρ περάσανε στο 50%. Επομένως η αγορά μπορεί να διευρυνθεί και μπορεί η διείσδυση των κοινοτικών στάνταρ σε άλλες χώρες να είναι πολύ μεγαλύτερη και εμείς θα δεσμευτούμε έτσι ώστε τα δικά μας στάνταρ να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και σε άλλες χώρες Λατινική Αμερική, στην Κίνα, στην Ινδία, σε όλες ε, τις αγορές ε, όπου το βιομηχανικό μας ε, σύστημα μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Τέλος, όπως σας είπα και στην ακρόαση, θα ξεκινήσουμε μια σειρά εντολών τυποποίησης, ας πούμε για την προστασία του καταναλωτού, για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουμε τη διαδικασία ε, αιτήματος ε, ε, προτύπου που συνδέονται με την οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Επίσης, να υπάρξουν περιβαλλοντικά στάνταρ και όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Τέλος, η προσβασιμότητα για αναπήρους και για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Το σλόγγαν είναι «Standard for all». Η τυποποίηση, όπως είπαμε και στην διάσκεψη World Standard Day, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στις πολιτικές προσβασιμότητας, κυρίως για ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού. Αρκεί να σκεφτούμε ότι περίπου ένα δέκατο ε, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει από κάποια μορφή αναπηρίας. Πρέπει, ε, ε, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι περίπου 10% της του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποια, ε, κάποιο πρόβλημα κινητικότητα. Ε, θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη ε, που έδειξε σε αυτό το τελευταίο σημείο, κυρίω μέσα από την υποβολή στην Ολομέλεια κάποιων τροπολογιών, οι οποίε οδηγούν ακριβώ σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό καταδεικνύει κατά πόσο γυτνιάζουν οι θέσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση της καινοτομίας, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, έχει αναφερθεί ε, κατά κόρο τον τελευταίο καιρό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εσωτερική μας αγορά βασίζεται σε ένα ευρύ δίκτυο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν ε, τεράστια πηγή θέσεων εργασίας, τεράστια πηγή απασχόλησης αλλά και ε, καινοτομίας ε, και που θα θέλουμε να αυξηθούν και στο μέλλον. Και βεβαίως μέσα και από τις αναδιαρθρώσεις των μεγάλων βιομηχανιών θα πρέπει να επανεστιάσουμε την προσοχή μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζεται η Small Business Act ε, έτσι ώστε να υπάρξει ένα στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς ενίσχυση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι νέες δράσεις της Small Business Act θέλουν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να έχουν αηφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τα θέματα τα οποία μας απασχολούν περισσότερο είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, τραπεζική πίστη, ε, η ενίσχυση της ένταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγορές που είναι όλο και πιο ε, διευρυμένες και παγκοσμιοποιημένες και βεβαίως να δώσουμε κίνητρα στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα και να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στην εσωτερική αγορά συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί έπαιξε πάρα πολύ και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, πρόθεση των δράσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίως βασίζομαι, υπολογίζω την στήριξή σας ε, για την ενίσχυση και την εφαρμογή ε, εφαρμογής της Small Business Act. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε ε, βάση της έγκρισης ε, της οδηγίας ε, για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αλλά βεβαίως τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει. Αυτό, αυτό το σημαντικό θέμα δεν έχει τελειώσει. Όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε πολύ μεταξύ ημών στην συνέντευξη τύπου. Τώρα πρέπει να περάσουμε στη φάση της ενσωμάτωσης, στη φάση της μεταφοράς. Και βεβαίως από κοντά θα παρακολουθούμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατάσταση. Πρέπει να περάσουμε λίγο τώρα στην ε, φάση της ε, ε, μεταφοράς και τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν ακόμα περισσότερο και βεβαίως καθόλου να μην χάσουν χρόνο στην εφαρμογή του κανονισμού που θα βάλουν σε κυκλοφορία 180 δις εκατομμύρια δίνοντας μεγάλη δόση οξυγόνου στις επιχειρήσεις μας. Χθες ε, το Κολέγιο των ε, Επιτρόπων συνάντησε τη μελλοντική Ουγγρική Προεδρία και ε, ζητήθηκε από την Προεδρία χωρίς καθυστέρηση και ανεπιφύλακτα να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στη Small Business Act και να εντάξει τα στοιχεία αυτά στα συμπεράσματα του Εαρινού Συμβουλίου. Επίση, και σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ε, να ε, ε, ευνοήσει την αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης που θα έχουν στη διάθεσή τους και για την ανάπτυξή τους οι επιχειρήσεις. Η δημιουργία, η ελεγχόμενη μάλλον εφαρμογή του μέσου εγγύησης για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει του καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας προχωράει με τρόπο αρκετά ικανοποιητικό. Μέχρι σήμερα έχουμε υπογράψει με διάφορους εταίρους 29 συμφωνίες βάσει των οποίων έχουμε ικανοποιήσει τις ανάγκες όσον αφορά τραπεζικό δανεισμό περισσότερων από 90.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ε, εγγύηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη φτάνει στα 200 εκατομμύρια ευρώ και μέσω της χρήσης του ε, θα ε, μέσω της χρήσης της μάλλον θα έχουμε ε, περίπου 7,5 δις ευρώ ε, δανείων ε, για τις επιχειρήσεις. Τώρα, το λέω και το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς καινοτομία. Ε, βεβαίως στη ανακοίνωση Ένωση για την Καινοτομία που ενεκρίθη στις 6 Οκτωβρίου είμαι βέβαιος το ελπίζω τουλάχιστον ότι θα φέρει ε, περαιτέρω απαντήσεις ε, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Ας πούμε θα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κεφαλαίου κινδύνου και την στρατηγική χρήση των δημοσίων διαγωνισμών. Επίσης και για να ε, μην υπάρξουν αρνητικές φορολογικές ε, ε, αντιμετωπίσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και θα προτείνει και μια νομική, νομοθετική συγγνώμη, πρωτοβουλία η οποία θα δημιουργήσει μια πραγματική εσωτερική αγορά του κεφαλαίου κινδύνου για τις εταιρείε, για τις επιχειρήσεις και για τους επενδυτές που θέλουν να καινοτομήσουν. Επίσης, η ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί στο ρόλο των δημοσίων διαγωνισμών, κυρίως δε των καινοτόμων, καθώς επίσης και των προ ε, εμπορικών ε, διαγωνισμών ε, που μπορούν να συμβάλλουν στην καινοτομία. Και όπως δείχνουν ήδη κάποιες εμπειρίες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτω χώρες, Φιλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία, αυτά τα εργαλεία τελικά αποδεικνύονται πολύ ωφέλιμα για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες μου αυτή τη στιγμή μελετούν ένα σχήμα και ένα μέσο χρηματοδότησης των των δημοσίων των ε, διαγωνισμών που αφορούν την ε, καινοτομία και επίσης υπάρχει μια γραμμή προπολισμού ε, για το θέμα αυτό για το 2011. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά τον τομέα των, της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γνωρίζετε ότι το 2010 ήταν έτος κλειδί για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είχαμε την έγκριση της ανακοίνωσης για τα καθαρά και οικολογικά οχήματα τα οποία το οποίο στηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, δημιουργήσαμε και την ομάδα υψηλού επίπεδου CARS 21. Ε, τέλος, ε, τη... Και τέλος είχαμε την πρόσφατη έγκριση των μέτρων συμμόρφωση για οχήματα έτσι ώστε να απλουστευτεί και να επικαιρωθεί επικαιροποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την έγκριση πολλών ε, μέσων εφαρμογής του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των ε, οχημάτων. Ε, είχαμε επίσης την έγκριση του νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τα τρακτέρ και επίσης είχαμε και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τυποποίηση των διτρόχων και τριτρόχων οχημάτων για το έτος 2011 ε, θα δεσμευτούμε έτσι ώστε ε, να περάσουν στη συναπόφαση αυτά τα μέτρα. Το 2011 επίσης ε, θα είναι έτος κλειδί για την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων όσον αφορά την τυποποίηση και την έρευνα υπέρ της πολιτικής προώθησης των πράσινων και ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2011 ε, θα εγκρίνει μια νομοθετική πρόταση για την ταξινόμηση των κρατών μελών που ήδη έχουν ταξινομηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Θα περάσω τώρα στην υφαντουργία. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς ε, για την εργασία που έκανε όσον αφορά ε, τον νέο ορισμό της υφαντουργίας. Περιμένουμε βεβαίω την κοινή θέση του Συμβουλίου γύρω στα τέλη του 2010. Στην κοινή θέση το Συμβούλιο θα πρέπει θεωρητικώς να, να εγκρίνει πολλέ από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Αλλά βεβαίω παραμένει ανοιχτό το ευαίσθητο πολιτικά ε, θέμα του σήματο προέλευση. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά το σήμα ε, προέλευση. Και όσον αφορά την, με την ευκαιρία μάλλον τη δεύτερη ανάγνωση, βεβαίω θα πρέπει να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσει έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Έχω ήδη συζητήσει με το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα το θέμα το οποίο πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περάσαμε από το επίπεδο κορεπέρα σε επίπεδο Υπουργών που νομίζω ότι έδωσε ε, και ε, ε, μεγαλύτερη πολιτική υφή και μεγαλύτερο πολιτικό βάρο στη θέση του Κοινοβουλίου. Και βεβαίω τι διεργασίε γνωρίζετε όλες, όλοι πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει λόγο να τι επαναλαμβανώ. Όσον αφορά τώρα τα, προϊόντα κατασκευή. Ε, ε, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να πω ότι πρέπει να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Στάιλερ γιατί οι προσπάθειές της σε αυτόν τον ιδιαίτερα περίπλοκο ε, τομέα ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται το μεγαλύτερο μέρος της πρότασής σας. Ας πούμε το κριτήριο της ανεξαρτησίας ε, που προτείνεται για τα σημεία επαφής των προϊόντων ε, μας φαίνεται πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την ανάγκη ε, εισαγωγής υποχρεωτικής δήλωσης για τις επικίνδυνες ουσίες, θα ήθελα να σας πω ότι ούτως ή άλλως στα πλαίσια του REACH υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση και νομίζω ότι θα πρέπει να καθησυχαστούν οι ανησυχίες σας. Επίσης, πρέπει να πω ότι δεν θέλουμε να βαρύνουμε ακόμα περισσότερο και ε, ε, με τρόπο εξαιρετικό ε, το βάρος το οποίο ήδη έχουν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην σημασία που έχει η πρόταση αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά πολυάριθμες στον τομέα της κατασκευής. Λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο, στο κανονιστικό κείμενο προβλέπει μία διάταξη οποία επιτρέπει στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, μια σχετική ευελιξία όσον αφορά τις διαδικασίες πιστοποίησης ε, των προτύπων, άρθρο 37 δίνουμε την ευκαιρία αυτή σε κάποιες πολύ μικρές επιχειρήσεις και αναφερόμαστε βεβαίως ε, σε κατηγορίες ε, προϊόντων που δεν προκαλούν προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων στα εργοτάξια. Ε, αυτό το μέτρο και νομίζω ότι καλό είναι να το υπογραμμίσουμε ορίστηκε στην πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την Better Regulation σαν ένα καλό παράδειγμα παράδειγμα εφαρμογής του Think First Principle, αυτής της αρχής, δηλαδή της πρώτης σκέψης. Τούτων ε, λεχθέντων ε, γνωρίζω ότι υπάρχουν στο, στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κάποιες διαφορετικές θέσεις όσον αφορά τα θέματα αυτά. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή με την στήριξη και του Συμβουλίου στο σημείο αυτό δεν είναι έτοιμη ας πούμε να, αφή, να δεν είναι έτοιμη να αφήσει κατά μέρος τις εξαιρέσεις για τις μικρομονάδες. Εν πάση περιπτώσει είμαι πεπισμένος πάντως ότι ότι ε, θα βρεθεί μια κοινή θέση την επόμενη εβδομάδα με το Κοινοβούλιο. Και ε, κύριε Πρόεδρε, ε, περαίνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βουλευτές που άκουσαν προσεκτικά και βεβαίως να υπογραμμίσω ότι με ενδιαφέρει να έχω μια καλή και στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η εργασία σας εδώ και ξέρω όμως και πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι για την καθημερινή ζωή της, των Ευρωπαίων πολιτών και εύχομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει όλο και πιο νομοθετικό ε, όργανο ε, και να είναι σε θέση να, να απαντά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα μελήματα των Ευρωπαϊκών πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, μια που ήταν πληρέστατη η εισήγησή σας, οι προτάσεις σας και οι ιδέες σας. Ε, αφορά μια τριετή περίοδο ε, η εισήγησή σας μια που αφορά την στρατηγική, το πρόγραμμά σας και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι τονίσατε θέματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή μας. Εποπτεία της αγοράς, ε, οδηγία για τα παιχνίδια, για παράδειγμα. Αυτό μας ενθαρρύνει ακριβώς όπως αφορά και τη δέσμη των μέτρων για τα εμπορεύματα, το ίδιο αφορά και του διαγωνισμού για το οποίο μιλήσατε και ο ίδιος έχω αναλάβει μια έκθεση ε, για το ζήτημα εκείνο και όσον αφορά την φαντουργία, πάλι και εκεί όπως ε, και για τα, τα μέτρα ε, που αφορούν τις ε, μετρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, εάν μπορείτε μείνετε μαζί μας μισή ώρα για να συζητήσουμε για να δούμε ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. σας θέλω το λόγο και εσείς, ναι, ναι, ναι, σας, ε, σας ανέφερα κύριε Ζουβά. E ε, Μιλήσατε κυρία, για το ΕΛΚ ή για δικό σου λογαριασμό ή για, για τον κύριο Σφάμπ. Έχετε το λόγο. Μαζί, μαζί. Χατσμπίλτ. Γκέπχαρτ. Mr. Trantafilides, Professor Correa de Campos, Mr. Juvin, Mr. Meyer and Mrs. Hanslick. Is everybody happy? Ε, αυτοί είναι οι αγορητέ. Είστε ικανοποιημένοι. Σα ε, ανέφερα όλου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για αυτήν την ανακοίνωση για την βιομηχανική πολιτική που καταδεικνύει την δέσμευση που έχετε αναλάβει απέναντι σε αυτή την Ευρώπη που διανύει σημαντικότατη κρίση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην πραγματική οικονομία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως τα εξής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, διακρίνουμε μία ε, απειλητική και επικίνδυνη αύξηση του προστατευτισμού ε, και ενώ εμείς θέλουμε καλύτερη κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά και αναφερθήκατε ας πούμε στα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν την είσοδο προϊόντων στη χώρα τους τους βάζοντας επιπλέον ε, προϋποθέσεις και στάνταρ και πρότυπα κτλ. Ε, επίσης ε, τον προηγούμενο Ιούνιο έγινε θεσμοθήκη το φόρουμ για την ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας. Εγώ είμαι η συγγήτρια για το θέμα αυτό και νομίζω ότι ε, έχοντας ε, μελετήσει πολύ το θέμα ε, με ενδιαφέρουν πολύ οι ορθές εμπορικές πρακτικές και τα private labels, οι ιδιωτικές ετικέτες που εφαρμόζουν πολλά σούπερ μάρκετ και διάφορες εταιρείες. Σας ρωτώ λοιπόν, προτίθεστε να κάνετε κάτι ε, ε, επιπλέον, ε, να προβλέψετε κάτι περισσότερο από την νομοθεσία η οποία ήδη υπάρχει και επίσης έχετε κάποια πρόθεση να κάνετε κάτι όσον αφορά τις σχέσεις B προς B μεταξύ επιχειρήσεων ο ίδιος ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε Ταγιάννη. Ήδη ανέφερα, δεν είχατε έρθει ακόμη, ότι ζητώ συγγνώμη εν ονόματι των άλλων μελών της πολιτικής μου ομάδος, διότι συνεδριάζουμε στην Βουδαπέστη. Εγώ έφυγα χθε το βράδυ και ήρθα για να παρίσταμε εδώ, αλλά αυτό εξηγεί γιατί είμαστε τόσο λίγοι σοσιαλδημοκράτες στη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ λέει ο επίτροπο. Δώσατε ε, μία σύντομη επισκόπηση πολλών πραγμάτων και δεν μπορώ στον περιορισμένο χρόνο να αναφερθώ σε όλα. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε τρία. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι τα άλλα είναι ε, πιο επουσιώδη αλλά δεν είναι δυνατόν να τα αναφέρω όλα. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι μία εισαγωγή η ε, deregulation, δηλαδή ε, η απελευθέρωση, αυτό μας έχει δείξει ότι μπορεί να οδηγήσει και σε καταστροφή. Οπότε απελευθέρωση δεν, μάλλον η ρύθμιση δεν σημαίνει προστατευσισμός, αλλά δίκαιος ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Αυτό επιζητούμε ε, στην πολιτική όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών και θέλω να το επαναλάβω για να μην υπάρχουν παρανοήσεις για την τοποθέτηση της πολιτικής μου ομάδος σε αυτό το θέμα. Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης ε, τι πιστεύετε σχετικά με το πρόγραμμα της ε, συνενώσεως, της συγκλήσεως των διαφόρων θεμάτων τα οποία αναφέρατε. Δηλαδή ε, στην θέματα που είναι τελείως διαφορετικά. Βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η συζήτηση ε, της ε, ε, οδηγίας των καταναλωτών όπου συγκεράζονται τέσσερις προηγούμενες οδηγίες. Είπατε λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε του χρόνου και σχετικά με μία απελευθέρωση δεν πρέπει να εκλειθούν θέματα τα οποία απλώς μπορεί να θεωρηθούν θεωρηθούν απλοποίηση. Υπάρχει μία οδηγία την οποία ανακαινήσαμε πρόσφατα και η οποία ακόμη εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Πριν λοιπόν να έχουμε μία εμπειρία σχετικά με τις καινοτομίες είναι σκόπιμο να υπάρξουν τροποποιήσεις και αναφέρομαι ε, στην πολιτική και την αλλαγή της έναντι των επιχειρήσεων και όχι μόνο των καταναλωτών. Ε, δεύτερο σημείο, εποπτεία της αγοράς. Πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική μας ομάδα και σήμερα πάλι με αυτά τα οποία είπατε ε, μου έκανε εντύπωση αυτό που αναφέρετε για τα προϊόντα τα οποία ήδη διατίθενται στο εμπόριο. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά στην αγορά και δεν αποσύρονται από την αγορά διότι για μας τους σοσιαλδημοκράτες η εποπτεία της αγοράς πρέπει να ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή ένα παιχνίδι που δεν είναι καλό για τα παιδιά δεν πρέπει καν να καταλήξει στο εμπόριο και θα πρέπει να φροντίσουμε τα, η οδηγία σχετικά με τα παιχνίδια να εφαρμοστεί σωστά στα κράτη-μέλη αλλά αυτό δεν μας επαρκεί στα κράτη-μέλη μας και υπάρχουν ακόμη οι κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν θέλει να ξανασκεφτεί τη θέση τη σχετικά με την ε, επιβεβαίωση των ε, πιστοποιητικών για τα παιχνίδια ιδίως για τα πολύ μικρά παιδιά που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ε, ήταν μια απέτηση ε, των σοσιαλιστών όπου δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε πλειοψηφία ούτε εις ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη τέτοια προϊόντα που κινούνται στην αγορά και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να μείνει το πράγμα έτσι. Και το τρίτο θέμα είναι η ε, σήμανση ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί των προϊόντων διότι αναφέρατε την ε, εκστρατεία πληροφόρησης. Την είχα παρακολουθήσει και πρέπει να σας πω ότι με ανησυχεί. Με ανησυχεί γιατί αυτή η εκστρατεία πληροφόρησης δίνει την εντύπωση στους πολίτες ότι ε, το δείγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ένα δείγμα ποιότητος, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές. Είναι ένα ε, σήμα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις και ε, το οποίο πιστοποιεί ότι συνάδουν και εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από τρίτους για να ε, υπάρξει επαλήθευση ότι πρόκειται για ασφαλή προϊόντα. Ε, δεν αναφέρεται όμως ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του σήματος, το CE. Εάν πώς, ε, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει να καταστεί ένα ε, ένα σήμα ποιότητος όπως ισχύει το αντίστοιχο σήμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποιήσεως το οποίο θα μας εξασφαλίσει ότι το κοινοτικό ποιοτικό είναι καλύτερο για να εγκαταλείψουμε τα εθνικά. Ε, και εγώ είμαι υπέρ της εναρμόνισης αλλά θα πρέπει να είναι μια εναρμόνιση ε, προς το καλύτερο. Αυτά είναι τα τρία σημεία τα οποία ήθελα να αναφέρω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, διμερώς ή κάπου αλλού, γιατί θέλω να αφήσω χρόνο και στους συναδέλφους να παρέμβουν. Ευχαριστώ κυρία Γκέφαρντ, ο κύριος Κρόισμαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, θα περιοριστώ σε δύο θέματα. Είπατε ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα και είπατε ότι ε, τα, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να κινηθούν σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αλλά έχω και μία άλλη ερώτηση. Κάνουμε αξιολογήσεις επιπτώσεων ε, που πρέπει να αξιολογήσουν και την περιβαλλοντολογική σκοπιά και την κοινωνική σκοπιά. Ε, πόσο αξιολογείται η ανταγωνιστικότητα και πώς ενσωματώνεται στα impact assessment διότι διαπιστώνουμε επανειλημμένως ότι από τη μία μεριά εμείς ε, λέμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί και από την άλλη πλευρά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, ε, ισχύουν οι ελάχιστες προδιαγραφές και όντως βλέπουμε στην εφαρμογή ότι υπάρχουν εμπόδια. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο μπορούμε να αντιπαραθέσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις στις μικρομεσαίες και πώς λειτουργούμε κοινωνικά. Και τέλος ε, είναι το θέμα της εποπτείας της αγοράς. Δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να υπάρχουν νέες ρυθμίσεις ε, αν δεν εφαρμόζονται. Ε, η εποπτεία όμως της αγοράς είναι θέμα των εθνικών κρατών και στη Γερμανία των γερμανικών κρατηδίων. Βλέπω λοιπόν ότι είναι δύσκολο να πληροφορηθώ για το πώς έχει το θέμα εφόσον μου λέγουν ότι στα κράτη-μέλη το θέμα της εποπτείας της αγοράς ρυθμίζεται τελείως διαφορετικά. Χρειάζεται και προσωπικό για την εποπτεία της αγοράς. Ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε, διότι πολλά από τα προϊόντα φτάνουν σε λιμάνια στην Ευρώπη και αν δεν έχουμε μία σωστή εποπτεία της αγοράς, τότε κυρία Γκέπχαρτ θα έχουν εισέλθει ήδη τα προϊόντα και δεν είναι δυνατόν λόγω της ποσότητάς τους να τα παρακολουθήσουμε. Επίσης ε, τι γίνεται με την συνεργασία παραδείγματο χάρη όσον αφορά την, ε, ε, την Frontex η οποία ασχολείται με την παράνομη μεταχείριση μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αρχές αυτές και στα λιμάνια και να εποπτεύουν την άφηξη των εμπορευμάτων ε, μπορούν να ε, υπάρχουν ε, να συστήματα όπως στην Αμερική που δεν αφήνουν να εισαχθεί κανένα προϊόν το οποίο έχει πιστοποιηθεί από μια τρίτη αρχή παρά μόνο αν έχει επαληθευτεί από Αμερικανική αρχή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να χειριστούμε και στον διατλαντικό διάλογο. Ο, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να πω ότι θα έρθει στην επόμενη συνεδρίαση και ο κύριος Ντεγκούχτ, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Εμπορίου, θα μπορείτε να του κάνετε παρεμφερείς ερωτήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολύ καιρό, θα παρακαλούσα να μην μακρηγορήσετε, ε, να περιορίσετε τις ε, παρατηρήσεις σας και να είστε λίγο πιο Κυρία Ρούλε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομη, έχω όμως τέσσερα και δεν νομίζω ότι πρέπει να πληρώσουν την ύφη τελευταίοι επειδή οι πρώτοι μακρηγόρησαν. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα κύριε Επίτροπε και βλέπετε ε, εφόσον έχετε ήδη εμπειρία σαν πρώην Ευρωβουλευτής ότι στο τέλος κάθε χρόνο ε, έχουμε ε, επικεφαλίδες στην εφημερίδα στη Γερμανία για τα παιχνίδια και τους κινδύνους. Βλέπουμε ότι το 80% των προϊόντων σε παιχνίδια που φτάνουν κάνει στην Ευρώπη δεν συνάδει με τη ρύθμιση περί της προστασίας των καταναλωτών. Ε, ζητάμε λοιπόν ε, για τα παιδιά να αγοράζονται κούκλες ε, από ύφασμα και όχι πλαστικές γιατί κινδυνεύουν τα παιδιά. Μου λέτε βέβαια ότι η οδηγία για τα παιδιά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να διευκρινίσουμε ποιε είναι οι αιτίες και γερμανική κοινή γνώμη θεωρεί ότι ευθύνεται η Ευρώπη. Μετά πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι οριακές τιμές για τα, προϊόν, για τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Πρέπει να εξετάσουμε και τις καρκινογόνες ουσίες. Αυτό που εγώ ζητώ είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια διότι όταν έχουμε έρευνες από διάφορα Ινστιτούτο θα πρέπει αμέσως να ενημερώνεται και το Ευρωκοινοβούλιο διότι ότι σε ε, την οδηγία για τα παιχνίδια είχαμε αναφερθεί και εις ε, την ε, ε, στον καθορισμό των οριακών τιμών για το θόρυβο στα πλαίσια της εναρμονήσεως και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν, ε, αν έχουμε τις πληροφορίες μπορούμε να επιδράσουμε καλύτερα και στην δημόσια γνώμη. Επίσης χρειάζεται καλύτερη εποπτεία. Υπάρχει ο κώδικας αλλά θα πρέπει να υπάρχει και παρκές προσωπικό κατά τρόπον ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σωστά. Αυτό όσον αφορά τα παιχνίδια, την εποπτεία της αγοράς πρέπει να συνεργαστούμε και μπορώ να διαβεβαιώσω την κυρία Κοράτσα Μπίλ ότι ε, δεν, ε, ε, δεν είμαστε υπέρ του προστατευτισμού αλλά αν είχατε στη χώρα σας επικεφαλίδες στις εφημερίδες ότι δεν καλύπτουν τις προδιογραφές τα παιχνίδια και εσείς θα, θα είχατε θορυβηθεί. Επίσης όσον αφορά τις ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιχειρήσεων και των καταναλωτών πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν αλλά θα περιμένουμε να δούμε το πακέτο που θα προτείνεται. Ε, όσο αναφορώ ε, το Small Business Act θα πρέπει να το αναβιώσουμε διότι πρέπει να δούμε και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει δηλαδή, δημόσιες προμήθειες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα και επίσης όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υποβολές ε, προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς θα είναι προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μπορεί να γίνει ε, μέσω του διαδικτύου διότι έχουμε άλλα προβλήματα όχι μόνο σαν ε, παραγωγή αλλά και σαν αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα και αν στηρίξετε μόνο τους βιομηχάνους θα πρέπει να ε, θα βλάπτονται οι ε, έμποροι και χρειάζεται μια συμβιβαστική λύση. Το θέμα αυτό είναι της ε, αρμοδιότητας του κυρίου Μπανιέ και υποθέτω ότι θα επανέλθει ο κύριος Μπανιέ σε αυτό. Ο κύριος Ρενταφυλίδης. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο κύριε Πρόεδρε, απλώς για να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Έχει κάνει αναφορά σε μια σειρά από δράσεις που προτίθεται να αναλάβει στο επόμενο διάστημα. Έκαμε αναφορά στην επιποπτεία της αγοράς, στην τυποποίηση των προϊόντων που είναι ζωτική σημασία για την προστασία των καταναλωτών που ιδιαίτερα ενδιαφέρει την δική μου ομάδα, αναφορά στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση της ε, καινοτομίας, όλα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ασφαλώς αντιλαμβάνομαι ότι αυτές είναι εξαγγελίες, έτσι την τελική μας κρίση θα την έχει όταν δούμε ότι όλα αυτά υλοποιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και πάμε τώρα στον ε, καθηγητή Κάμπος και κατόπιν οι υπόλοιποι, οι καθηγήτρια, οι Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας επισκεφθήκατε. Όχι, ο κύριος Κάμπος, ο καθηγητής Κάμπος έπρεπε να λάβει το λόγο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και ξαναπαίρνει το λόγο. Δεν κατάλαβα καλά. Σε ποιον δώσατε το λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι με μεγάλη μας χαρά σας ακούσαμε κύριε Επίτροπε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί το έργο σας τα απαιτεί αυτά. Για να μπορέσετε να πετύχετε όλους αυτούς τους στόχους που έχετε τάξει. Έχουμε το θέμα της ε, οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές. Έχουμε επίσης και τη συμβάση μεταξύ επιχειρήσεων, που είναι ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί. Οπότε, για πέστε μας για ε, τα ζητήματα αυτά. Τι μπορείτε να κάνετε ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να μην αργούν να εφαρμόσουν τις οδηγίες γιατί τα νομοθετήματα που σας ανέφερα τα χρειάζονται οι επιχειρήσεις, ιδίως τώρα που περνάμε αυτή την κρίση. Επομένως θα πρέπει πριν περάσει η διετία να έχουν εφαρμοστεί τα προαναφερθέντα μέτρα. Μήπως μπορείτε με δύο λόγια να μας πείτε τι ισχύει όσον αφορά τα οχήματα τα οποία Ήδη έχουν βγάλει πινακίδε σε ένα κράτο μέλο και κανεί θέλει να αλλάξει χώρα. με αυτό γίνεται αυτό, να βγάλουν πινακίδε αλλού. Πώ μπορεί κανεί να εκμεταλλευτεί την ε, κινητικότητα και να δουλέψει σε χώρα προέλευση, σε χώρα διαφορετική συγγνώμη από τη χώρα προέλευσή του. Εγώ φταίω, εγώ φταίω, λέει ο πρόεδρο. Δεν ήμουν σαφή στην έδωσα το λόγο τώρα τον δίνω στον καθηγητή Κάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Εσείς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εσείς διαλέξατε κάποια θέματα να μας τα παρουσιάσετε. Θεωρήσατε ότι αυτά μας ε, ενδιαφέρουν. Εμείς σας ακούσαμε και θεωρήσαμε ότι με το συγκεκριμένο σας χαρτοφυλάκιο ε, μπορείτε να καλύψετε και ζητήματα πέραν της εσωτερικής αγοράς. Και εσείς επομένως έρχεται να μας πείτε αυτό το οποίο νομίζετε ότι θέλουμε και εμείς σας ε, ρωτούμε αυτά τα οποία θέλουμε πραγματικά να μάθουμε τέλος πάντων. Ε, με φιλικό τρόπο μπορεί αυτό το προβληματάκι να ξεπεραστεί και να δούμε ας πούμε τι γίνεται όσον αφορά τα μέτρα, τα εποπτικά για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα. Νομίζω ότι τα μέτρα, τα προτινόμενα είναι τα κατάλληλα ε, όσον αφορά και αγαθά και υπηρεσίες. Ε, αναφερθήκατε και στο παράδειγμα της Ρωσίας, πάνε εύστοχο και είμαι στη θέση να σας πω ότι συμφωνούμε με τα περισσότερο μας είπατε όσον αφορά την χρηματοδότηση της πολιτικής καινοτομίας. Τώρα όσον αφορά την εσωτερική αγορά, τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ε, πάρα πολύ ωραία, τα είπατε. Όμως, για πέστε μας, όλα αυτά τα ωραία πράγματα πώς θα υλοποιηθούν. Εσείς είστε και αντιπρόεδρος της Επιτροπής και μας εξηγήσατε το νομοθετικό ε, πρόγραμμα, το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για του χρόνου Και όταν διαβάζω τι προβλέπεται για την ιστορική αγορά, εκπλήσωμαι. Διότι εσείς θα πρέπει να πείτε στους 12 συναρμόδιους συναδέλφους σας να τους πείτε ποια είναι τα προβλήματά μας, ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν εδώ. Τι γίνεται με την πρωτοβουλία Μόντι. Έχει ξεφουσκώσει. Κατέληξε όλη αυτή η υπόθεση σε αυτά τα έξι μέτρα που εδώ αναφέρεται για την ενιαία αγορά. Αυτό με τίποτα δεν είναι η υλοποίηση της ενιαίας πράξης. Αισθανόμαστε απογοήτευση λοιπόν. Ευχαριστούμε καθηγητή Κάμπος. Κύριε Ζουβέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε επίτροπε, να σας πω κάτι το οποίο χτες το άκουσα την εξής ιστορία. Το εξής περιστατικό. Και ίσως δεν είναι καν απλό περιστατικό, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Μου το είπε ένας ε, ε, κατασκευαστής αναπτύρες αν κατασκευάζει τόσο πίσω που μου το είπε, πολύ σημαντικός και ε, δρά εδώ στην Ευρώπη είπε επομένω ότι 70% των αναπτύρων που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Κινέζοι προέρχονται από την Κίνα γιατί οι αναπτύρες όπως είπατε κι εσείς, διέπονται από κάποιες προδιαγραφές. Και 70%, 76% των εισαγωμένων και πολλουμένων στην Ένωση δεν ε, ανταποκρίνονται σε αυτές τις προδιαγραφές, όμως έχουν το σήμα σε κάτι το οποίο μας οδηγεί σε 40 νεκρούς ετησίως λόγω της κακής ποιότητας αυτών των αναπτύρων. Όμως έχει και αποτελέσματα οικονομικά αυτή η κατάσταση, διότι σε μια δεκαετία από το 100% που είχαμε που κατασκευαζόντουσαν ε, εδώ, έχουμε μόνο 30% των πολλωμένων που κατασκευάζονται στην Ένωση. Άρα έχουμε σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Άρα τι διαπιστώνουμε. Επιβάλλουμε προδιαγραφές, όμως Υπάρχει συμμόρφωση και γιατί όχι. Θα πρέπει πρώτα πρώτα του κανόνες να του εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές. Γιατί πολλές φορές παρά είναι οικείς. Και από ό,τι μου είπαν υπάρχει κάποια ε, υπηρεσία. Ας πούμε η υπηρεσία μου είπανε του λιμένους του Ρότερνταμ δεν λειτουργεί όπως πρέπει και γι' αυτό και έχει πλημμυρίσει η Ευρώπη από τέτοια προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνουν με τις προδιαγραφές μας. Επίσης είναι απίστευτο το ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε αγορές εκτός Ευρώπης. Σε αγορές όπως της Βορειοαμερικής όπου υπάρχει συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Άρα, αρκεί κανείς να θεσπίζει τέτοιες διατάξεις ή θα πρέπει να φροντίζει και για τη συμμορφωσή τους ακόμα και από τις εθνικές υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τους αναπλήρες. Είμαι σίγουρος και άλλα προϊόντα. Εμφανίζουν τα ίδια αποτελέσματα και όλα αυτά φυσικά θα τα πούμε την Πέμπτη στις 18. Οπότε την Πέμπτη τέλο πάντων όταν θα σας πω πότε είναι ακριβώς θα έρθει ο κύριος Ντεχούχτ. Κύριε Μάιρ Ευχαριστώ. Συμφωνώ σε πολλά θέματα με τους συναδέλφους, γι' αυτό και θα παραμείνω σε δύο θέματα, στα δομικά υλικά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν θέσεις εργασίας, θέσεις εκπαίδευσης και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις αυτές να μπορούν να χρησιμοποιούν και κεφάλαια υψηλού κινδύνου πρέπει να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση της κοινή αγοράς διότι βλέπουμε ότι ε, έχει σημασία να υπάρχει ε, και η σωστή σήμανση. Θέλω να μιλήσω όμως και για τις μικροεπιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις ε, ως προς την αδειοδότηση και ούτω καθεξής και πρέπει να πω ότι εγώ είμαι ε, περισσότερο όλο και πιο πολύ προπομπός της ε, απελευθερώσεως και κατά της γραφειοκρατίας. Βλέπω όμως ότι στη Γερμανία χρειάστηκε να ε, περιορίσουμε πολλά πράγματα κατά τρόπον ώστε το Ινστιτούτο των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικροεπιχειρήσεων να μην τύχει εκμεταλλεύσεως και πρέπει το να ε, ε, επιδιορθώσουμε την κατάσταση. Διότι ζητήσαμε με τους συναδέλφους να διαγραφεί αυτή, αυτές ε, οι έκτακτες διατάξεις και είμαι έτοιμος προς συμβιβασμό όπως και, και οι συνάδελφοι αλλά για ποιο λόγο. Όπως σας είπα ο περιορισμός αυτός, οι περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν στη Γερμανία έχουν κοινοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέμε δηλαδή μικρο, ε, μικρο επιχειρήσεις μέχρι 9 ε, εργαζομένους και 2 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Πρέπει να γνωρίζει κανείς πώς διαχωρίζονται από τις τεράστιες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν μια στρατιά μικροεπιχειρήσεων για να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει επανόρθωση και ε, να διορθωθεί, να αποκατασταθεί η κατάσταση και θα περιοριστώ σε αυτό και στην αίτηση την οποία διατύπωσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε συνάδελφοι πάρα πολύ ενδιαφέρουσαν η ανταλλαγή των απόψεων και όπως καταλαβαίνετε κύριε Επίτροπε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο σας από, από πολλές οπτικές γωνίες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι τις εξελίξεις μαζί και όλα αυτά που είπατε θα τα συνεχίσουμε εμείς να τα συζητάμε εσείς βέβαια πρέπει να φύγετε αν μπορείτε απαντήστε σε όσα μπορείτε όσο μπορείτε θα σας, ε, σας ευχαριστώ και θα δώσω σύντομες απαντήσεις. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο είδα να αναδύεται είναι το θέμα της εποπτείας της αγοράς. Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που ακούστηκαν επί του θέματος αυτού που καταδεικνύει βεβαίως τη σημασία που του αποδίδεται. Και είναι ένα θέμα στο οποίο είναι πολύ ευαισθητοποιημένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή μου δεν τίθεται το ζήτημα με όρους ε, εποπτεία έναντι προστατευτισμού. Ε, κάποιοι κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται δεν είναι απαραίτητο ότι θεσπίζονται για να προστατευτεί κάποιο εθνικό συμφέρον. Εγώ πιστεύω ότι σωστές εθνικές ρυθμίσεις, σωστοί εθνικοί κανόνες ε, απλώς προστατεύουν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Ε, με την προϋπόθεση βεβαίως να μην θέλουν να κλείσουν ακόμα περισσότερο την αγορά, αλλά να θέλουν αντιθέτως να την ε, ανοίξουν. και βεβαίως και με την προϋπόθεση οι κανόνες οι εθνικοί αυτοί να μην αντιτίθενται ε, στους κανόνες που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως, εγώ αναφέρθηκα στην καλύτερη διακυβέρνηση και απαντώ εδώ στην κυρία Γκέμπχαρτ. Βεβαίως η better regulation θα πρέπει εφιώς να υλοποιηθεί. Θα πρέπει να βοηθήσουμε στην απλούστευση των διαδικασιών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιο εύκολα ε, τους ε, κανόνες, ε, να διασφαλίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ακριβώς ε, και απαντώ και στον κύριο Κρόσμαν, όταν μιλάω για ανταγωνιστικότητα, ε, και γιατί τη συνδέω με την Better Regulation. Εμείς έχουμε αναφέρει στην ανακοίνωση για την μηχανική πολιτική μία σειρά ε, δοκιμασιών, τεστ ανταγωνιστικότητας. Όλες οι ρυθμίσεις που προτείνουμε στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο πριν βγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει επιτυχώς μια δοκιμασία αξιολόγησης ανταγωνιστικότητας. Ένα τεστ, όχι όμως που θα γίνεται μονάχα εξάντε εκ των προτέρων, αλλά και εξπόστο εκ των υστέρων. Όταν δηλαδή αρχίσει να ε, εφαρμόζεται ε, ο κανόνας σε ένα υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεν, θα, δεν αρκεί να μην αντιτίθεται στην ανταγωνιστικότητα, αλλά το σύνολο του συστήματος θα πρέπει να συντονίζεται με τις δράσεις υπέρ της ε, ανταγωνιστικότητας. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Επίσης, Έχουμε εισαγάγει την ιδέα ενός κειμένου για την ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις διεθνείς ε, εμπορικές συμφωνίες. Δηλαδή, πριν υπογραφεί οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα ή όχι της συμφωνίας αυτής επί της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιριών. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει ανακοίνωση στο Συμβούλιο ε, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων βιομηχανικών τομέων ε, και την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση μονάχα ελέγχοντας το ε, δημόσιο χρέος, που βεβαίως είναι απαραίτητο και αυτό, αλλά και μέσω της αύξησης της ανάπτυξης και της εποπτείας της εσωτερικής αγοράς. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία, αυτό είναι πολύ ευρύ θέμα βεβαίως και περιλαμβάνει και την εφαρμογή του σήματος ΣΥΗ. Εγώ δεν τροποποίησα τις επιλογές του προκατόχου μου κυρίου Φερχόγγεν. αλλά βεβαίως είμαι πρόθυμος να συζητήσω οποιασδήποτε υπόνοιε ή οποιασδήποτε αμφιβολίε. και ευχαριστώ και την ε, κυρία Γκέπχαρτ γιατί μου έδωσε τροφή προσκέψη. Είναι σαφές ότι όλοι θέλουμε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι και το είπα και στην ε, ακρόαση απαντώντας την ερώτηση ενός ε, συναδέλφου σας, του κυρίου Πιτέλα, ο οποίος είναι επόμενη σήμερα και ο οποίος αναφέρθηκε ακριβώς στο σήμα CE και στο σήμα ποιότητος. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σήμα ποιότητα τα επόμενα χρόνια, αλλά και ε, σε σχέση και με αυτά που λέγατε κι εσείς, ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε σωστά το ε, σήμα ΣΥΗ και όχι εναλλακτικά ε, με άλλα σήματα τα οποία κάποιες χώρες ενδεχομένως χρησιμοποιούν και που βεβαίως μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει αντίθεση εδώ. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε σωστά το σήμα CE, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ συχνά υπάρχουν απάτες όσον αφορά την χρήση του σήματος CE. Ε, ε, ε, το ξέρουμε αυτό και επομένως πρέπει να λάβουμε και τα μέτρα μας. Γιατί κάθε φορά που βλέπουμε ένα προϊόν με το σήμα CE δεν είναι απαραίτητο ότι το προϊόν αυτό πραγματικά έχει περάσει όλο τον έλεγχο των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σήμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν αφορά σήμα ποιότητος, είναι ένα σήμα τυποποίησης και πάντως χρειαζόμαστε χρόνο. Εποπτεία της αγοράς. Ένα θέμα το οποίο πολλοί μεταξύ ημών έθεσαν. Εγώ μίλησα με κάποιες αποχρώσεις. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπωσδήποτε θέλει και προτίθεται να σεβαστεί την αρχή της επικουρικότητας. Εμείς δεν έχουμε ε, δυνατότητα αστυνομικού ελέγχου είτε στα σύνορα είτε στους εσωτερικών των χωρών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε σωστούς κανόνες, να έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα υποπτίας, να επιμείνουμε ε, στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τους ε, κοινοτικούς ελέγχους είναι γεγονός αυτό που, που αναφέρατε ότι σε κάποιους λιμένες δεν εφαρμόζεται σωστά ο έλεγχος. Μα προς τα εκεί θα πάνε οι προσπάθειές μας ε, ε, και βεβαίως εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε και όσον αφορά την κατάρτιση των ελεγχόντων. Αυτοί που κάνουν τους ελέγχους θα πρέπει να είναι καλά καταρτισμένοι, να ξέρουν αν υπάρχει καταχρηστική χρήση του σήματος ή εάν τα ε, προϊόντα, κυρίως δε τα παιχνίδια εάν ελέγχονται με σωστό ε, τρόπο. Να σας πω ότι στη χώρα μου πριν από δύο-τρεις μέρες κατασχέθηκαν ε, ε, χιλιάδες χιλιάδων κινέζικης προέλευσης παιχνίδια τα οποία δεν ανταποκρίνονται εις, τις, στα ευρωπαϊκά πρότυπα κατασκευής και τα κατάσχεσε λοιπόν η αστυνομία όλα αυτά τα παιχνίδια. Ε, θα πρέπει λοιπόν η έλεγχη να είναι σαφής, αυστηρή, διαρκής ε, σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου και στα τελωνία και στις, ε, στα χερσαία σύνορα και στους λιμένες έτσι ώστε να ξέρουμε εάν τα προϊόντα είναι επικίνδυνα, αν είναι παραχαραγμένα κτλ. Όσον αφορά την οδηγία για τα παιχνίδια γνωρίζουμε ότι ε, βεβαίως ε, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ε, ενός ε, κανόνα μπορεί αυτός να χρειαστεί να αλλάξει. Το γνωρίζουμε αυτό και βεβαίως κατά περίπτωση θα αξιολογούμε τα διάφορα στοιχεία και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίοι αξιολογούν και στα πλαίσια του ΡΙΤΣ και βάσει της επιτροπολογίας ε, διάφορες κυρίως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, για τις αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες και βεβαίως εμείς θα κινηθούμε βάσει των κανόνων και φυσικά εγώ δεσμεύομαι να μεταδώσω, να μεταφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα στοιχεία τούτων ελεγχθέντων και όσον αφορά πάντα την εποπτεία των αγορών και θα σας απαντήσω στα γαλλικά. Έχουμε ήδη την ε, ε, διάταξη για την ε, ενιαία εφαρμογή του 765. Έπειτα έχουμε και ένα πλαίσιο για την διεύρυνση του απέξε του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκυρης Ειδοποίησης. Επίσης έχουμε την οδηγία για τα προϊόντα, τα κοινά προϊόντα συχνής χρήσης Βεβαίως υπάρχουν και τα εθνικά προγράμματα εποπτείας και πρόγραμμα ελέγχου από τα τελωνία. Βεβαίως τα κράτη-μέλη μας έχουν απαντήσει, έχουν δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας ε, των αγορών και μας έχουν δώσει και τον κατάλογο των ε, υπηρεσιών ελέγχου και εποπτείας. Φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και την συνεργασία μας με την Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική, Αμερική και Καναδά. Dans les marchés E Επιστρέφω στα Ιταλικά. Όσον αφορά την πρόσβαση ε, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους ε, δημόσιους ε, διαγωνισμούς, βεβαίως θέλουμε η πρόσβαση αυτή να είναι απρόσκοπτη. Ε, θέλουμε οι εταιρείε, οι επιχειρήσει αυτέ ε, όχι μονάχα να έχουν πρόσβαση στου διαγωνισμού αυτού, αλλά να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την επιχειρηματική και εμπορική ζωή των χωρών. Ε, είναι σαφή ο ρόλο που θα παίξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εσωτερικής αγορά της Ιδία αλλά θα πρέπει να δούμε και τη σημασία και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπό το φως και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις μεγάλες ε, βιομηχανίες. Εμείς δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας σε μία επιχείρηση. Εμείς πρέπει να στηρίξουμε την απασχόληση και νομίζουμε ότι ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν πηγή ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας η, θέλουμε να προστατέψουμε την αγορά, όχι την αγορά για την αγορά, αλλά την αγορά σαν ένα εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει, σαν ένα μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε στον προβληματισμό των πολιτών, σαν ένα μέσο να απαντήσουμε ε, στα προβλήματα των πολιτών. Σχετικά με την ερώτηση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ ε, για την διατροφική αλυσίδα. Ναι, υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της την προηγούμενη εβδομάδα στην ομάδα υψηλού επίπεδου εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς από τον γεωργικό μέχρι ε, τους ε, τελικούς ε, καταναλωτές. Εκπροσωπούνται μάλιστα και εταιρεί, συγγνώμη, φορείς προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων. Επομένως, στην ομάδα αυτή θα υπάρχουν οι γεωργοί, θα υπάρχουν οι προστάτες των δικαιωμάτων των ζώων, θα υπάρχουν οι προστάτες ε, των ε, καταναλωτών και Και γνωρίζετε βεβαίως ότι στην κοινή γεωργική πολιτική ε, και στο πρόγραμμα το οποίο μόλις εγκρίναμε και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό ακριβώς εγώ καθυστέρησα γιατί είχαμε έτσι μια επιμήκυνση της ε, ε, συζήτησης ε, γιατί μιλούσαμε ακριβώς για προτάσεις που αφορούν την κοινή γεωργική πολιτική και μάλιστα λέγω ότι σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της συζήτησης για την κοινή γεωργική πολιτική και με, την, με τις λιανικές πωλήσει. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ και λέγω ότι όντως προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή όχι μονάχα τους επιτρόπους, όχι μονάχα τους βουλευτές αλλά και εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων μερών και μάλιστα έχω συζητήσει και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ ο οποίος ε, συμφωνεί να ε, ε, συζητηθεί και το ενδεχόμενο ένταξης νέων ε, ρυθμίσεων. Ε, εγώ δεν αποκλείω κάτι τέτοιο, όπως δεν αποκλείω ε, και στη διάρκεια των συζητήσεων να υπάρξουν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα προσπαθήσουν, θα προσπαθήσουν να καλύψουν προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν στη διάρκεια της συζήτησης για τη διαδροφική αλυσίδα. Όσον αφορά τώρα τα, την αυτοκίνητο βιομηχανία και τα αυτοκίνητα. Ακόμα κάνουμε impact assessment. Δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα μια ε, πλήρη ε, και ενδελεχή απάντηση. Δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα διορθώσουμε το τελικό ε, κείμενο. Όσον αφορά την εποπτεία, απήντησε και προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάποιες ε, παρατηρήσεις σε αυτά που είπε ο καθηγητής Κάμπος. έχει υποβληθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας οδηγήσει προς την πράξη για την εσωτερική αγορά Internal Market Act. Και δεν υπάρχει μονάχα το κείμενο του Μάριο Μόντι. Μπορούμε να είμαστε βεβαίω όλο και πιο φιλόδοξοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε θέση να μετατρέψουμε σε πράξεις και σε ρυθμίσεις κάποιες ε, ε, προτάσεις και όσο πιο φιλόδοξες τόσο πιο δύσκολο να υλοποιηθούν. Βεβαίως ο καθένας μας έχει κάποιες πολιτικές ε, πρωτοβουλίες, ο καθένας μας έχει κάποιες πολιτικές φιλοδοξίες και νομίζω ότι στα λεγόμενά σας ο κύριος Μπαρνιέ έχει ήδη εν μέρει απαντήσει στα μελήματα τα οποία εκφράσατε έχει ήδη εν μέρει απαντήσει ο κύριος Μπαρνιέ και ο οποίος επίσης έχει μια μακρά ε, πείρα ως βουλευτής και επομένως γνωρίζω ότι σέβεται, και θα σέβεται το Κοινοβούλιο και θα ανταποκριθεί στα αιτήματα αιτήματά του. Όσον αφορά τώρα τα υλικά κατασκευών, τα δομικά υλικά, ε, θεωρώ ότι, και το είπα και προηγουμένως, ότι μπορεί να εξευρεθεί ε, συμβιβασμός όσον αφορά τις μικροοντότητες, τις μικροεπιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή στις προτάσεις και τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχοντας όμως, διατηρώντας όμως κάποιες ε, επιφυλάξεις και κάποιους προβληματισμούς. Πάντως είμαι απολύτως ε, διατεθειμένος να συζητήσω ανοιχτά ε, και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο που όμως θα στηρίζει και τις μικρές και ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις γιατί επαναλαμβάνω είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, και στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση της καθυστέρησης πληρωμών είμαι απολύτως διατεθειμένος να συζητήσω ε, το θέμα. Υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες ήδη ισχύουν κάποιες ε, ρυθμίσεις και που πρόλαβαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως εμείς θα ζητήσουμε από όλες τις χώρες ε, μέλη να κινηθούν γρήγορα. Αλλά η πρότασή μας μπορεί να είναι μονάχα πολιτικού χαρακτήρα. Δεν μπορούμε ε, να επέμβουμε ε, με άλλο τρόπο Ελπίζω και ευελπιστώ όλοι να κινηθούν ε, γρήγορα. Το, βεβαίως ε, λόγω προβλημάτων οικονομικών, λόγω ε, ψηλού χρέους ενδεχομένως κάποιες χώρες να τροποποιήσουν την αντιμετώπιση τους αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με όλα αυτά τα, τα στοιχεία μπορούν οι χώρες να βγουν μία ώρα αρχίτερα, μία ώρα νωρίτερα από την κρίση την οποία οποία να διανύουν. Και συμφωνώ απολύτως, μια και μιλάμε για δημόσιο χρέος, συμφωνώ ότι δεν αρκεί μέσω μειώσεων κλπ. κλπ να ε, ε, μηδενίσουμε το δημόσιο χρέος. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ταυτόχρονη ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και από την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και πολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμές ευχαριστίες με εξ όλων για την πλήρη παρουσίαση αλλά και για το ότι απαντήσατε σε τόσες πολλές ερωτήσεις τόσο καλά και στην εισήγησή μου σας είπα ότι εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεργασία μαζί σας και στον επόμενο κύκλο που θα νομοθετήσουμε θα συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο Οπότε επίσης θα είναι χρήσιμο για το θετικό πνεύμα των υπηρεσιών συνεργατών σας αλλά και ότι προσωπικά ενδιαφέρεστε για όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε και μείνατε τόσο πολύ. Αν ασχοληθήκατε με τόσα πρακτικά θέματα, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συμμετέσχουν στη συζήτηση. Γκέμπχαρτ και Κάμπος, ιδίως αυτούς τους συναδέλφους ευχαριστούμε που ήρθαν για αυτή τη συζήτηση εδώ για να μπορέσουν να βοηθήσουν ε, ε, από πλευρά απόψεων των πολιτικών του ομάδων και εδώ τελειώνει η σημερινή μα συνάντηση, συναδέλφοι, αλλά θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, σα υπενθυμίζω. 7 και 4 για να ψηφίσουμε σε αυτή την οδηγία τα προϊόντα κατασκευών. Ε, ο κύριο Μάγερ έχει θέματα να μα αναπτύξει εκεί. Επίση, στι Βρυξέλλε θα συνδέουμε στι 29 ενδεκάτου τη Δευτέρα στις 3 η ώρα. Οπότε θα έχουμε τον συνάδελφο του κ. Δαγέννη, τον κύριο Φούχτ, για κάποια ζητήματα εμπορική πολιτικής.